Συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε. Κύριε Βαντενκάμπ, σας περιμένουμε. Με την άνεσή σας. Όλα έτσι κι αλλιώς στην ώρα τους θα γίνουν με την άνεσή μας. Στην υγειά σας κύριε Βαντενκάμπ. Νομίζω ότι το σημερινό απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενο και αν όχι απλώς ενδιαφέρον, σίγουρα συναρπαστικό. Θα ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση με ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές μας ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, με την κυρία Κάρλα Πέις δηλαδή και τον κύριο Μπράιαν Σίμψον που γνωρίζουν πολύ καλά την Επιτροπή αυτή. Περιμένω. Κύριε Σίμψον, ξέρετε πολύ καλά την Επιτροπή αυτή, έτσι δεν είναι. Μας γνωρίζετε. Στην ε, ανταλλαγή αυτή θα ασχοληθούμε με το θέμα της πολυδιαλογικότητας, με, τους, με τις λεωφόρους της θάλασσας, και την ε, πρόοδο του διαδρόμου Ρήνου Δούναβη. Περιμένουμε πολλά από εσά, κύριε Σίμψον. Θα σας προσέχουμε με τεντωμένα τα αυτιά. Και μετά θα ακούσουμε και τους συντονιστές μας που θα μας κάνουν την τιμή να έρθουν, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν κάπως την κατάσταση και μετά τους συντονιστές της δικής μας επιτροπής τον κύριο Πίπερ και τον κύριο Ερτούκ. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα σας ακούσουμε πολύ προσεκτικά και μετά θα σας θέσουμε ερωτήσεις γιατί είμαστε γεμάτοι περιέργεια. Λοιπόν, κυρία Πέις, σας δίνω το λόγο ιδίως για αυτό το θέμα που μας ενδιαφέρει. Πώς θα ασχοληθούμε με την πολυδιαλογικότητα και πώς προχωρά ο διάδρομος Ρήνου Δούναβη. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητή Καρύμα, αν με επιτρέπετε, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να σας παρουσιάσω το θέμα αυτό της πολυδιαθρολογικότητας και της σχετικής διοργάνωσης όπως παρουσιάζεται στο πρόσφατο έγγραφο ο συνδυασμό των διαφόρων μέσων μεταφορά, η πολυδιαλογικότητα, λόγω χάρη συνδυασμό ναυσιπλοεία και σιδηροδρόμων, είναι και το αντικείμενο τη Λευκή Βίβλου του 2011 για να καθορίσουμε και μια σχετική ε, πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Εδώ ασχολούμαστε με διαδρόμους, ε, με πολυδιαλογικά μέσα μεταφοράς, ώστε να αξιοποιήσουμε όλα τα συστήματα πληροφορικής, ε, τη λογιστική που διαθέτουμε και τη μεταφορά εμπορευμάτων ε, σε όλο το μήκος των διαδρόμων. Και προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες ευρωπαϊκές ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις για να έχουμε και την κατάλληλη εφοδιαστική μέρημνα. Εδώ είχαμε και μια σχετική ανταλλαγή υπόψεων με τους υπευθύνους από τον Μάρτιο. Θα σας εξηγήσω γιατί οι Ευρωπαίοι συντονιστές αποφάσισαν να ασχοληθούν γεωγραφικά με τους διαφόρους διαδρόμους, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και κάποια οριζόντια ζητήματα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες που έχουν σχέση με την πολυγεωλογικότητα που σχετίζονται με τα δίκτυα μεταφοράς. διότι τα, η αστική κόμβη είναι κάτι κοινό μεταξύ όλων των διαδρόμων έτσι κι αλλιώς, αλλά η αντιμετώπιση και η κάλυψη αυτών των θεμάτων είναι σημαντική για το δίκτυο συγκοινωνιών τη Ευρώπη και για να αντιμετωπίσουμε και του στόχου ε, των κλιματικών αλλαγών. Θα επικεντρωθούμε εδώ στις ευφυεί και αποτελεσματικές λύσεις μεταφορών, αλλά όλο ιδιαίτερος στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε με τον καλύτερο τρόπο ε, να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη των δικτύων αυτών σε συνδυασμό με τις επενδύσεις. Πώς μπορούμε να ε, συνδυάσουμε τα πολυδιαλογικά συστήματα, ιδίως τους σιδηροδρόμους και τις αυσιπλοείες και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις Πώς τις υλικέ εγκαταστάσεις και τις ευφύ εγκαταστάσεις μπορούμε να τις διασυνδέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να έχουμε καλέ υπηρεσίες εφοδιαστικής είναι μια σημαντική διάσταση ώστε οι μεταφορές να γίνουν πιο βιώσιμες και να μειώσουμε και το αποτύπωμα άνθρακα αναπτύσσοντας την αγορά. Στο σχετικό έγγραφο είχαμε ορίσει κάποιες ανάγκες επενδύσεων για τις πολυγελογικές μεταφορές καθώς και την εφοδιαστική για τους διαδρόμους με το εμπόριο με σχετικούς στόχους. Οι επενδύσεις βάσει των κυρίως δικτύων θα πρέπει να ε, στοχεύσουν καλύτερα τι διάφορε προοπτικέ του κάθε διαδρόμου. Και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στι επενδύσει, ε, στι πλατφόρμε εφοδιαστική και στου κόμβου των δικτύων ε, συγκοινωνία. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν τοπικά και περιφερειακά προγράμματα που να διαχειριστούμε με την κατάλληλη διακυβέρνηση για τα, για τα σωστά αποτελέσματα. Θα πρέπει να υπάρξουν οι σωστές διασυνδέσεις των ε, υποδομών για να έχουμε αποτελεσματική εφοδιαστική. Θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες εμπορευμάτων και να λάβουμε υπόψη και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Γνωρίζω και είμαι ικανοποιημένη που η Επιτροπή αυτή έχει κάνει ήδη την ε, ε, δουλειά της για το θέμα αυτό και ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Γιάλα Σέντερ για την έκθεσή της. Συμφωνούμε σε πολλά σημεία μαζί σα, όπω για τον καθοριστικό ρόλο τη εσωτερική ναυσιπλοεία και των σχετικών διαδρόμων, ω μέσου για να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση τη αφοδιαστική. Επίση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει τη ψηφιοποίηση ή τι μοναδικέ προκλήσει τη απαλλαγή από τον άνθρακα. Ο διάδρομο Ρήνου Δούναβη συνδέει εσωτερικέ χώρε τη Ευρώπη, την, την Γαλλία, την ε, Γερμανία, την Αυστρία, την ε, Δημοκρατία τη Τσεχία, την Ουγγαρία, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Για να μην μιλήσω για χώρε που είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Σερβία. Πριν φτάσει να εκβάλει στον εύξηνο πόντο. Μιλάμε για 6.000 ε, χιλιόμετρα μήκο. 5.000 χιλιόμετρα δρόμων και 3.500 εσωτερικής ναυσιπλοείας που περνούν από 9 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και 4 μη ευρωπαϊκά ε, κράτη-μέλη. Χώρες που δεν είναι μέλη δηλαδή. Μιλάμε για δύο θαλάσσια λιμάνια, 14 λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοείας και 27 σταθμούς που ασχολούνται μόνο με το, που είναι μόνο ε, χρήσης. Η διευκόλυνση για την διασύνδεση της Ευρώπης έχει ε, βελτιώσει τους στόχους πράσινης οικονομίας και τους περιβαλλοντικούς φιλικούς ε, πολυδιαλογικούς τρόπους με εκατοντάδες προγράμματα ανά την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει σε πραγματικά έργα και αυτό έγινε ιδίως μεταξύ 2014-2015 με 14,5 ε, δις ευρώ να έχουν προβλεφθεί από το ΣΕΦ ως σήμερα. Είναι 2,2 τα δις ευρώ που έχουν προβλεφθεί για τους πολυδιαλογικούς τρόπους με 57 ε, δράσεις για το συγκεκριμένο διάδρομο και περίπου 3 τα δις για ένα μέρος του διαδρόμου μερικά παραδείγματα για το πώς η πολυδιαλογικότητα και η σχετική διαχείριση της εφοδιστικής έχουν αναπτυχθεί στο διάδρομο Ρήνου Δούναβη. Ο διάδρομος αυτός έχει σχέση με το πλωτό του Δούναβη. Και τα διάφορα μέσα κοινωνία έχουν να κάνουν με τις βιώσιμες και θεμετές συνθήκες ανταγωνισμού. Η ανακαίνιση του διαδρόμου αυτού έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη, η οποία συντονίζεται από, τα Ρουμανικά, από το Ρουμανικό και Αυστριακό Υπουργείο Μεταφορών. Το τελευταίο πρόγραμμα έχει εντοπίσει όλες τις τοποθεσίες όπου χρειάζονται βραχυπρόθεσμα μέτρα για να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει η σωστή ε, αναμόρφωση και εκμετάλλευση των πόρων. Θα πρέπει επίσης να εντοπιστούν σωστά τα προβλήματα και να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα βλέπουμε την αφοσίωση των μεγαλύτερων περισσότερων από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη να ε, δώσουν περισσότερε εγκαταστάσει για την εσωτερική ναυσιπλοεία το 2014. Και υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να ενώσουν τι δυνάμει του για την ε, καλύτερη εκμετάλλευση του Δούναβη. Η συνεργασία έγινε όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά εκφράστηκε και σε ένα κοινό πρόγραμμα του ΣΕΦ που ονομάζεται Fairway Danube με τη συνεργασία 6 χωρών Αυστρία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Το πρόγραμμα αυτό βασίστηκε σε εθνικά προγράμματα δράσης που καταρτίζονται δύση και ένα εργαλείο παρακολούθησης. Τον Μάιο του 2016 επικαιροποιήθηκε εν ώψη της συνάντησης των Υπουργών Μεταφορών στο Ρότερνταμ στις 20 Ιουνίου 2016. Ε, το πρόγραμμα αυτό συζητήθηκε για δύο μέρε και ε, παρατηρήθηκε πώς έχουν εκπληρωθεί οι δεσμεύσει του 2014. Υπάρχει όχι μόνο ένα γενικότερο πρόγραμμα, αλλά και τα πρώτα βήματα στην πράξη. Έχουν καταγραφεί τα στοιχεία για την κήτη του ποταμού, ε, μετρήσεις για τα περιβαλλοντικά και στοιχεία για την ναυσιπλοεία, για τα σκάφη και για, το, για τους εργαζομένους. Επίσης, και για οι εγκαταστάσεις για τις φορτηγίδες θα εγκατασταθούν ως νούπο ε, στον διάδρομο αυτό. Ως προς το νέο σκάφος ελέγχου της Κροατίας, θα έχουμε την τιμή να το βαφτίσουμε τον Οκτώβριο του 2017 στο Βούκοβαρ. Εδώ θα δείτε τους 37 τερματικούς σταθμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στα πλαίσια του διαδρόμου αυτού ορεινού Δούναβη. Μεταξύ άλλων και για τα ε, σκάφη μετρήσεων. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα της χρηματοδότησης. Υπάρχει η πρόκληση να συνδυάσουμε εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ώστε να μπορούμε να υλοποιήσουμε προγράμματα για την σωστή ανάπτυξη του διαδρόμου, η Βουλγαρία λόγω χάρη. Με το γενικό πρόγραμμα ε, εντοπίζεται ότι δεν έχει αρκετά σκάφη παραγλώδησης, περιπολικά. Θα πρέπει επίση να δούμε τα λειτουργικά προγράμματα για τι μεταφορέ και τι υποδομέ μεταφορών από το 2014 έω το 2020. Γιατί μπορέσαμε και στο Ρους να ε, βαφτίσουμε το σκάφος Midmarch με τον ίδιο σκοπό στο επίπεδο τη Βουλγαρία ενίσχυση των εγκαταστάσεων τη εφοδιαστική επιτρέπει την καλύτερη διασύνδεση των συστημάτων πληροφοριών για την ανταλλαγή δεδομένων και ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τη λογιστική και τη εφοδιαστική σε δύο τομεί. Πρώτον, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθου. Και δεύτερον, τη βελτιστοποίηση τη ε, μετακίνηση, τη μεταφορά των φορτίων και τη εκμετάλλευση όλων των εγκαταστάσεων. Μια ε, καλύτερη συνεργασία και συνεργασία το των απαιτείται και οι χώρε που έχουν το μέγιστο συμφέρον εδώ να αναλάβουν περισσότερε δραστηριότητε. Η εφοδιαστική και η συνδυασμένη πολυδιαλογικότητα μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε καλύτερα τι προσπάθειε μεταφορών εμπορευμάτων ώστε να χρησιμοποιείται καλύτερα το σύστημα μεταφοράς, ε, μεταφορών. Ε, εμπορευμάτων. Το σύστημα πληροφορική και οι τεχνολογικέ λύσει πρέπει επίση να αξιοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική ναυσιπλοεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τι υπηρεσίε πληροφοριών που διαθέτουμε. 15 εταίρια από 13 ευρωπαϊκέ χώρε έχουν ενώσει τι δυνάμει του σε όλη την Ευρώπη για να προχωρήσουμε στο, στην προσπάθεια αυτή ώστε να υπάρχει διαρκής προσφορά ε, πληροφοριών για τις ε, μεταφορές στο επίπεδο της ναυσιπλοείας και των σιδηροδρόμων με ένα κοινό πρόγραμμα. Το βασικό στοιχείο αυτού του συνδυασμού είναι όλοι οι εταίροι τη εσωτερική ναυσιπλοείας και των σιδηροδρόμων που χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε μέσω της πληροφορικής, να ε, ανταλλάσσουν με το βέλτιστο τρόπο της πληροφορίας για να διαμορφώνεται το καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για του λιμένες ελπίζουμε σε αύξηση τη αποτελεσματικότητα των μεταφορών τη εσωτερική ναυσιπλοεία. Με καλύτερη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, τη μείωση του χρόνου αναμονή και των διαδρομών, τη άρση των διοικητικών ε, φραγμών και την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων σκαφών. Είχα την τιμή να εγκαινιάσω την πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Λιμένων στο Βερολίνο τον ε, Ιανουάριο του 2017. Η πολύ διαλογική, εφοδιαστική, απαιτεί ισχυρά μέσα συγκοινωνιών, καλές εγκαταστάσεις, σωστά τοποθετημένε. σε κομβικά σημεία, όπως οι λιμένε, οι λιμένες εσωτερική οι πλατφόρμες εφοδιαστική, τα αστικά κέντρα και ούτω καθεξής, με καλά εργαλεία πρόσβαση. τα πολυδιαλογικά μέσα μεταφορέ πρέπει να είναι διασυνδεμένα σωστά και ψηφιακά και υλικά. Εδώ απαιτούνται στοχευμένες επενδύσεις σε εφικτά σχέδια με υποδομές στα κατάλληλα κομβικά σημεία. Επίσης, απαιτείται η κατάλληλη ψηφιακή πρικοδότη του συστήματος με διαλογικότητα και διαλειτουργικότητα. Λόγω χάρη στο διάδρομο που προανέφερα, το λιμάνι του Γιώργιου είναι ένα χαρακτηριστικό πράσινο λιμάνι που έχει πετύχει κάποιο από αυτού του στόχου. Πρώτα απ' όλα απαιτείται μελέτη και μετά η υλοποίηση των έργων. Η μελέτη εδώ ξεκίνησε το 2012. Για να έχουμε την σωστή τεχνική ανάλυση και να έχουμε μια καινοτόμα απόκριση στις ανάγκες των λιμένων, Στο Γιώργιο συγκεκριμένα μπόρεσε να αναμορφωθεί και να αξιοποιηθεί καλύτερα το λιμάνι με τη συμμετοχή τοπικών εταίρων. Τους ίδιους τους χρήστες και τον ίδιο το βιομηχανικό κλάδο που θέλησε να αξιοποιηθεί αυτός ε, ο διάδρομος. Το ε, έργο αυτό στηρίχθηκε από το ΣΕΦ το 2014 στο επίπεδο της συνοχής. Η διαχείριση του έργου και η επικοινωνία ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία. Μετά περάσαμε στη φάση της οικοδόμησης με ένα ε, τριπλό σύστημα μέσων μεταφοράς συνδυασμό οδικών, ε, σιδηροδρομικών και πλωτών δρόμων. Επίσης για να πάρει την πιστοποίηση του περιβαλλοντική της περιβαλλοντικής ε, συμμόρφωσης στο λιμάνι αυτό, ανέλαβε τα κατάλληλα μέτρα. Ναι. Το ε, θέμα της γεωγραφικής διάστασης του διαδρόμου Ρήνου Δούναβη ε, Ω προ τη διαλειτουργικότητα και τη διαλογικότητα των βιώσιμων συστημάτων μεταφορά στην περιοχή έχει καθοριστική σημασία. Οι οδικέ και οι σιδηροδρομικές μεταφορέ πρέπει να διαχειριστούν καλύτερα και για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και των επιφατών. Οι ε, μεταφορέ εσωτερική ναυσιπλοεία μπορεί να δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα και να επιτρέψουν ευρύτερη ανάπτυξη όλη τη περιοχή. Βεβαίω το αν θα προχωρήσουμε, όλα αυτά εξαρτώνται από την πολιτική βούληση να αναπτυχθεί αυτό ο διάδρομο. Πρέπει να υπάρξει βιώσιμη και αξιόπιστη διαχείριση με τα κατάλληλα κριτήρια. Θα πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσει στην εσωτερική ναυσιπλοεία και τι εγκαταστάσει τη, μειώνοντα το κόστο των μεταφορών. Συμπέρασμα. Πολλά έχουν γίνει, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ακόμη συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου για την τρίτη γενιά των σχετικών προγραμμάτων που αναμένουμε γύρω στο 2018. Ωστόσο, τα προγράμματα εργασίας μετά την ανάλυση των εγκαταστάσεων διαδρόμου είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να ολοκληρώσουμε τις φιλοδοξίες μας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στο 2030. Η πρώτη φάση του σχεδίου ε, ήδη έχει καθυστερήσει. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, τα ξέρετε από τις χώρες σας φαντάζομαι. Γι' αυτό παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την ε, ολοκλήρωση του βασικού δικτύου. Σε στενή συνεργασία με τα κάτι μελη τους διαχειριστές των υποδομών και όλους τους εταίρους των διαδρόμων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλα τα διασυνοριακά προγράμματα. Για να αποφύγουμε τα σημεία συμφόρησης θα πρέπει να δούμε τις οριζόντιες προτεραιότητές μας, οι οποίες θα πρέπει να αναπτύσσονται πλήρως πολυδιαλογικά και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πολιτικές πτυχές, ε, όπως η καινοτομία, τα εναλλακτικά καύσιμα, η ασφαλή στάθμευση και το καθεξής. Μόνο με αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση, οι διάδρομοι θα ικανοποιήσουν τις επιθυμίες και προσδοκίες των πολιτών και των ε, εταιριών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κυρία Πέις. Κάρλα με λένε. Κάρλα. Αν μου επιτρέπετε να σας ε, αποκαλώ Κάρλα. Ευχαριστώ πολύ για την τόσο εξαντλητική και λεπτομερή παρουσίαση. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον κύριο Μπράιν Σίμψον που θα εστιάσει σε ένα θέμα το οποίο ε, ενδιαφέρει πολύ κόσμο και είναι έτσι αναδυόμενο. Είναι η περίφημες θαλάσσιες Έχετε ένα τέταρτο παρακαλώ για την παρουσίαση αυτή Σα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και μέλη τη Επιτροπή Χαίρομαι που ξαναγυρίσα και πάλι στην Επιτροπή μας. Την τελευταία φορά που είχα έρθει ήταν πέρσι τον Ιούνιο, όπου παρουσίασα το πρώτο πρόγραμμα εργασίας για το μέλλον των θαλασσίων λεωφόρων και ελπίζω σήμερα να έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε. Το 2017 είναι θαλάσσια χρονιά, είναι εντατική συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων στην ναυτιλία για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση για το πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία και για την Ευρώπη και να ε, αναθεωρήσουμε και να εξυγχρονίσουμε ε, το θεσμικό πλαίσιο στη ψηφιακή εποχή για τις θαλάσσιες μεταφορές. Μετά την αρχική παρουσίαση της Κάρλα Πέις, θα ήθελα να σας πω πόσο σημαντική είναι η πολιτική των θαλασσίων λεωφόρων γενικότερα στους διαδρόμους των μεταφορών. Είναι μια οριζόντια εγκάρσια προτεραιότητα των διευρωπαϊκών δικτύων δεν εννοείται ένα δίκτυο μεταφορών ενιαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συστήματα συνδυασμένων μεταφορών. Χάρη στις θαλάσσιες λεωφόρους ε, έχουμε 40% του εσωτερικού εμπορίου και 75% του εξωτερικού και στους ευρωπαϊκούς λιμένες φτάνουν αγαθά που δεν σταματούν εκεί, αλλάζουν το μέσο μεταφοράς και ε, παραδίδονται στο βάθος της ενδοχώρας στον τελικό πελάτη. Συνδέονται λοιπόν οι θαλάσσιες λεωφόροι και το βασικό δίκτυο ε, των διαδρόμων και είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε πραγματικά να αποδώσουν αυτά τα δίκτυα. Στα πλαίσια όλων αυτών πρόσφατα ε, εγκρίθηκε αντίστοιχη δήλωση στη Βαλέτα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολιτική υποστήριξη και βόληση από πλευράς κρατών μελών έτσι ώστε να έχουμε διαδρόμους για συνδυασμένες μεταφορές, για μεταφόρτωση με νέες ε, τεχνολογίες, νέες εγκαταστάσεις και αποτελεσματική όσο και βιώσιμη υποδομή. Επίσης με χαρά διαπίστωσα ότι έγινε ρητή αναφορά στην ε, κρίσιμη συνεισφορά των κατευθυντήριων γραμμών των ε, ευρωπαϊκών δικτύων και της ε, διευκόλυνσης στην Ευρώπη. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε ε, πάνω από 80 τακτικά δρομολόγια από πάνω από 400 λιμάνια που συνδέονται παγκοσμίως. Τρία από τα 29 λιμάνια αναφέρονται ε, στην, ε, στους αντίστοιχους κανονισμούς και 79 θαλάσσιοι λιμένες βρίσκονται ε, στην άκρη ενός από τους εννέα βασικούς διαδρόμους, κεντρικούς διαδρόμους. Αυτό σημαίνει τα δύο τρίτα της συνολικής ε, κίνησης των ευρωπαϊκών λιμένων. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο ε, με τις μεταφορές, είναι και κλάστερ εφοδιαστικής και βιομηχανίας που δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας. Πέρσι τον Ιούνιο σας παρουσίασα το πρώτο πρόγραμμα δράσης μου ε, σε λεπτομέρειες. Το κείμενο βασίζεται ε, σε τρεις πυλώνες ε, της ναυτιλίας που έχω θεωρήσει έχω προτεραιότητες. Σας θυμίζω λίγο ποιοι είναι αυτοί. Το πρώτος είναι το περιβάλλον. Μπορούν οι θαλάσσιες φόροι να βοηθήσουν τον κλάδο να τηρούν την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία του Διεθνούς Οργανισμού Αυτά έχουν να κάνουν με την ποιότητα του αέρα και ε, τον έλεγχο των εκπομπών θείου. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται και ε, ε, τα εναλλακτικά καύσιμα όπως είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, για αποθήκευση και τερματικά LNG, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τη ρήπανση από την αυτιλία, από τη λειτουργία. Το δεύτερο βασικό που έχουμε στόχο είναι η ένταξη ε, στις αλυσίδες ε, εφοδιαστικής των ε, θαλάσσιων μεταφορών. Ναυτιλία δηλαδή και λιμενικές υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορούν να δοθούν και στη θάλασσα και στη στεριά. Η ψηφιοποίηση μπορεί να κάνει τα συστήματα μεταφορών να είναι πιο αποτελεσματικά και να οδηγήσει σε καλύτερη χρήση υφισταμένων πόρων και υποδομών. Επίσης μπορεί να μειώσει το ε, γραφειοκρατικό άκθος, ε, να βελτιώσει τη διαχείριση ε, της προσφοράς και να αυξήσει γενικά την απόδοση των μεταφορών και της λογιστική, συγγνώμη. Το 2015 η Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ δημιούργησε ένα φόρουμ, ένα συμβουλευτικό όργανο, μια πλατφόρμα για το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων στις συνδυασμένε μεταφορές. Και διακλαδικά, ένα από τους βασικούς στόχους του φόρουμ είναι να ε, είναι πιο εύκολη η ε, ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών στο περιθώριο των διαδρόμων. Σήμερα ε, οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών ε, λειτουργούν ε, σε σύλλο απομονωμένοι χωρίς να διασυνδέονται και να ανταλλάσσουν προφορίες. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί και να έχει μια οριζόντια κάθε διάταξη. Αυτές τις προτεραιότητες ε, χρηματοδοτούμε ε, έργα που ε, αυξάνουν τη σύνδεση της ναυτιλίας με την παράκτια αλία στην Ευρώπη, το short shipping, τεχνολογίες πληροφορίας, επικοινωνίας με συστήματα διαλειτουργικά και συγκεκριμένες δράσεις καλύτερες συνδέσεις με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές θα πρέπει επίσης να ε, αυξάνει η χωρητικότητα και ενδεχομένω να υπάρχουν και επεκτάσεις όπου χρειάζεται. Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι ιδιαίτερα. Το σύστημα της παγκόσμιας, διαχείρισης παγκόσμιας κίνηση, κίνησης έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν ε, οι ε, κυκλοφορίες και οι ροές των φορτίων σε φορτηγά Επίσης, ε, υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο και η κατάρτιση. Αυτό μιλάει από μόνο του. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, κατάρτιση νέες τεχνολογίες, όπως ε, διαδικασίες ε, αποθήκευσης LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλα. Πώς κατανέμεται ο προϋπολογισμός που έχουμε για τις θαλάσσιες λεωφόρους. Μέχρι τώρα είναι 651 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό θα επικεντρωθώ τα δύο τελευταία χρόνια στο ΣΕΦ, Connecting Europe. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει επιχορηγήσεις 360 εκατομμύρια ευρώ που ε, πήγαν σε 40 ευρωπαϊκά έργα και συνολικά ε, προσέλκυσαν επενδύσεις ε, της τάξης των 965 εκατομμυρίων ευρώ. Τα περισσότερα χρήματα δαπανήθηκαν σε έργα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε LNG, σε ε, διάφορα συστήματα υποδομών ε, που να είναι συμβατά με το ΣΕΚΑ, πιλωτικά προγράμματα, ηλεκτρικά σκάφη και ε, διάφορα συστήματα παροχής προσφοράς onshore στη ξύρα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για το περιβάλλον. Blue Baltics, η γαλάζια Βαλτική. Αυτό βοηθάει ε, να εφαρμοστούν οι κανονισμοί ΣΕΚΑ και ΜΑΡΠΟΛ ε, με ένα καθαρό καύσιμο που είναι το ε, υγραέριο ε, για τους ενδιαφερομένους. Το project αυτό είχε μία δράση στην Λιθωνία και στην Εστονία και Στόχος είναι να διερευνηθεί η ε, χρήση ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλτική για τις μεταφορές. Τούτο λεχθέντων δεν θέλω να αφήσω να δημιουργηθεί εντύπωση ότι υποστηρίζουμε μόνο το υγραέριο. Ε, στην πολιτική μας γενικά υποστηρίζουμε τα εναλλακτικά καύσιμα και τις αντίστοιχες υποδομές. Αυτό φαίνεται από ένα άλλο έργο που υποστηρίζει τη μεθανόλη και πάλι από τα αντιευρωπαϊκά δίκτυα, που είναι το ε, θαλάσσιο καύσιμο του μέλλοντος. Υπάρχει ένα φεριμπότ που λέγεται στένα Τζερμάνικα και με κάποιες ε, προσαρμογές και ανακατασκευές ε, δοκιμάζουμε τις αποδόσεις που έχει με τη μεθανόλη. Επίσης, οι διατροπικές ε, συνδυασμένες μεταφορές ε, συνδέομαστε και με το Ισραήλ για ένα διάδρομο για την ε, κυκλοφορία νοπών τροφίμων. Αυτό έχει να κάνει με κοντέινερ που, από όπου μεταφέρονται από το Ισραήλ ευαλείωτα τρόφιμα προς ε, διάφορα λιμάνια, μεταξύ αυτών ε, στη ε, Μασαλία. Φως. Κερδίζουμε χρόνο, βοηθούμε το περιβάλλον και υποστηρίζουμε και τις συνδυασμένες μεταφορές. Τέλος, η πρόταση και η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά ένα άλλο ενδιαφέρον έργο που είναι η διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας. 12 κρατημέλη υπό την αιγίδα των Σουηδών συμμετέχουν σε ένα έργο που έχει 42 εκατομμύρια προϋπολογισμό για ε, τυποποιημένη ε, πληροφόρηση, ανταλλαγή πληροφοριών, εξετάζει τον ε, διάπλου και τις αφήξεις στα λιμάνια και παρέχει όλες τις βασικές ε, υπηρεσίες. Διαχείριση των ροών, ε, συστήματα συνεργατικά για λήψη αποφάσεων και διαχείριση πληροφοριών. Είναι και πολύ μεγάλο το δυναμικό, 12% μείωση ε, καυσίμου, μείωση του χρόνου ελιμενισμού και κινητοποίηση στα λιμάνια, αγκυροβόλησης και γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σύστημα STM ε, για τη διαχείριση της θαλάσσιας ε, κυκλοφορίας ε, εμπορευμάτων θα είναι επαναστατικό και θα θέσει τα ορόσημα για τις εισαγωγές και εξαγωγές. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το STM είναι συμβατό επίσης με την ενιαία θηρίδα για τη θάλασσα, την οποία θα προτείνει το χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στα πλαίσια αυτά, επίσης, θα παρέχουμε και το σκέλος που αφορά τη θάλασσα για τους ε, διαδρόμους συνδυασμένων μεταφορών ε, στην ε, ψηφιακή ατζέντα και στο φόρουμ για την εφοδιαστική. Τώρα, από εδώ και μπρος τι γίνεται. Από την περσινή μου παρουσίαση άρχισα μια διαδικασία διαβούλευσης με κράτη-μέλη και τους ενδιαφερομένους από τον κλάδο με τον εξή στόχο. Να συζητήσουμε το μέλλον της πολιτικής των θαλασσίων λεωφόρων που είναι από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος εργασίας μας. Ο τελικός στόχος είναι να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του και να είναι πιο ειδικό και να δούμε ποιες είναι εκείνες ε, οι ε, πολιτικές που είναι πιο κρίσιμες για το μέλλον. Θα σας αναφέρω και τους πυλώνες για την ανάπτυξη, αλλά ε, επικεντρώσουμε στο περιβάλλον, ας πούμε, θα πρέπει να εστιάσουμε στη, στα εναλλακτικά καύσιμα. ή όταν μιλάμε για την αλυσίδα εφοδιαστικής χρειάζεται περισσότερη προσοχή ε, στην σύνδεση με το, τις θαλάσσιες λεωφόρους ή να δούμε κάποια άλλα στοιχεία. Όταν όταν μιλάμε για την βελτιστοποίηση της μεταφοράς φορτίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, στη διαχείριση των θαλασσίων ροών ή να εστιάσουμε περισσότερο στην κατάρτιση και στα εναλλακτικά καύσιμα. Όλα αυτά είναι ερωτήσεις και ερωτήματα που τίθενται. Και ε, το τελευταίο εξάμεινο έχω λάβει πάρα πολλά ε, σχόλια, ε, απαντήσεις ε, από λιμενικές αρχές, από εφοπλιστικές εταιρείες, από διαφέρους ενδιαφερομένους. Και φέτος θα έχω ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο ε, εργασιών και πρόγραμμα εργασιών που θα δημοσιευθεί. Είναι αδιαμφισβήτητη υποστήριξη των λεωφόρων της θάλασσας και γενικώ θεωρείται ότι θα πρέπει να περιορίζεται σε συγκεκριμένα ε, έργα για τη χρηματοδότηση και να αντανακλά καλύτερα τις συζητήσεις που γίνονται ε, στο φόρουμ για τη βιώσιμη ε, αλία και το άλλο φόρουμ για την εφοδιαστική και τις μεταφορές. Θα πρέπει να συνδυαστεί όλο αυτό με τους κάθετους διαδρόμους μεταφορών για να δούμε πώς θα συνδυάσουμε καλύτερα τη φιλοδοξία των θαλασσίων λεωφόρων με τις γενικότερους στόχους. Ορισμένοι λέγουν ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα 29 λιμάνια ή να είμαστε πιο επιλεκτικοί στις δράσεις μας. Οι λεωφόροι αυτοί να, αυτές να είναι η σύνδεση με τα νέα κεντρικά διευρωπαϊκά δίκτυα. Μια άλλη λύση είναι να έχουμε ένα συνολικό δίκτυο λεωφόρων για όλους τους λιμένες. Ε, το σημερινό μέγεθος των πλοίων μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση ε, φορτίου ε, στους μεγάλους λιμένες και αυτό να είναι προς μειονέκτημα των μικρών. Υποστηρίζουμε κάθε δράση που βοηθάει στο πρασίνισμα του ευρωπαϊκού στόλου για να τηρείται περισσότερο και πιο αυστηρά η περιβαλλοντική νομοθεσία, να έχουμε νέες υποδομές για τα νέα καύσιμα, να αφήσουμε να βοηθήσουμε τη Βαλτική να χρησιμοποιήσει νέα καύσιμα και να περιορίσουμε τη ρήπανση γενικότερα. Για την περιφέρεια, τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, γίνεται ευρύτερη συζήτηση για το πώς θα γίνονται καλύτερες διασυνδέσεις με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Πέρα από τη χρηματοδότηση, ε, από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο λόγω της γεωγραφικής τους ε, απομόνωσης και θέσεις. Εγώ είμαι σε στενή επαφή πάντα με τα κράτη-μέλη και τους ενεχορμένους για να ε, δούμε πώς μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις θαλάσσιες λεωφόρους και αυτές οι πρωτοβουλίες. Για μένα είναι κρίσιμο να εξασφαλίσουμε η πολιτική των θαλασσίων λεωφόρων ανακλάται και σε πολιτικές προτεραιότητες και ε, την αντίστοιχη χρηματική ε, πρικοδότηση. Ε, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική η χρηματοδότηση με επιχορηγήσεις από το Connecting Europe. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κλάδος, να καινοτομεί και να βρει νέες λύσεις για να είναι πιο πράσινη η λειτουργία, πιο αποτελεσματική και πιο καθαρή. Ζητώ την υποστήριξή σας και για το πρόγραμμα δράσης και γενικότερα για τις αλλασίες λεωφόρους όταν θα έρθει η στιγμή να αρχίσετε να συζητάτε για τον προπολογισμό. Ε, είμαστε λίγο το αποπέδι της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών ε, ενώ θέλω πραγματικά να γίνουμε αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σίμψον για την παρουσίαση αυτή και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σμελ Ερτούγκ που είναι και ένας από τους μόνιμους εισηγητές για το θέμα αυτό. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω εδώ, dear Brian. Αγαπητέ Brian, καλώς ήρθες στο Κοινοβούλιο. Δύο θέματα έχω να σχολιάσω. Το πρώτο είναι ότι δεν γνωρίζω αν η σημασία του MOS είναι γνωστή στα κράτη-μέλη. Και... Των θαλάσσιων λεωφόρων δηλαδή. Το πιο σημαντικό εμπόδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε τους στόχους που ανέφερες είναι πολύ γνωστό και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ήταν οι καθαρές μεταφορές που συζητήσαμε, το σχετικό κανονισμό. Μια οδηγία συγκεκριμένα πάρα πολύ σημαντική. Ίσως η πιο καλά προετοιμασμένη οδηγία της Κομισιόν. Έπειτα βέβαια είχαμε την εξή κατάσταση. Τα κράτη-μέλη και ιδίως το δικό μου, αλλά και άλλα, βλόκαναν την κατάσταση και τώρα δεν έχουμε ποσοτικά μέτρα, ούτε στόχους. Και τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να έχουν υποβληθεί νομίζω μέχρι τα τέλη, έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2016. Αλλά τα περιμένουμε αυτά τα εθνικά σχέδια δράση και από ό,τι άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5-6 κράτη-μέλη έχουν στείλει ήδη τα εθνικά σχέδια δράση του στην Κομισιόν. Αν το συγκρίνουμε αυτό με του βασικού σα στόχου. Μα εξηγήσατε και πάρα πολύ σωστά τα λέτε, ρο, ρο, CNG, λιμάνια κτλ. Πώς εντάσσονται όλα αυτά πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας όταν τα κράτη-μέλη... Δεν ξέρω πώς να, τους χαρα... να τα χαρακτηρίσω, δεν σπάω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι απρόθυμα, ας πω, αυτή την ε, έκφραση να χρησιμοποιήσω. Πώς μπορούμε να τα πιέσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δουλειά τους. Να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Τουλάχιστον έστω να καταρτήσουν τα εθνικά σχέδια δράσης. Και το δεύτερο θέμα, που είναι και ένα ερώτημα, η Επιτροπή Μεταφορών, εμείς δηλαδή, νομίζω ότι πριν από τρεις μήνες είχαμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια αποστολή στη Γαλλία. Και επισκεφτήκαμε και το λιμάνι της Μασαλίας μεταξύ άλλων, όπου για πρώτη φορά, είμαι ειλικρινής και το παραδέχομαι, ότι ήταν η πρώτη φορά που άκουσα κι εγώ, που υπήρχε αυτός ο διάδρομος ε, για τα φρέσκα φρούτα, για τα νοπά ε, φρούτα. Πρώτη φορά το άκουγα, ήταν συζήτηση αυτό. Όταν ε, μιλάμε για αυτή την εισαγωγή αυτών των νοπών φρούτων από το Ισραήλ, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα θαλάσσιας αρτηρίας αυτό. Πώς θα πετύχαινε όμως αν δεν συμπεριλαμβάνονταν οι περιφερειακοί φορείς. Ξέρουν έχουν ενημερωθεί ότι κάτι σχεδιάζεται. Δεν νομίζω. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε ως συντονιστής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μπορεί να κάνει για να διαδώσει καλύτερα στους περιφερειακούς φορείς αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε. Και ένα άλλο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη που κάποιες φορές ε, δεν μετακινούνται Για να δω τον κατάλογό μου. Ο Βιν Βαντενκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ακούσαμε τη λέξη Brexit καθόλου. Γιατί ήταν η πρώτη ερώτησή μου. Σίγουρα προς τον Brian Simpson. Και τώρα τι θα γίνει με τις θαλάσσιες λεωφόρους σε σχέση με σε σύνδεση ή ρήξη της σύνδεσης με τον Brexit. Είναι ο τέταρτος γύρος αυτός που έχουμε με τους συντονιστές των ε, διαδρόμων, ε, των διευρωπαϊκών. Το μοντέλο που προτείνουν οι ε, συντονιστές και τη γενική τους εισαγωγή το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Όλοι οι συντονιστές δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, αλλά μεταξύ τους ασύνδετη και ασυντόνιστοι, Ενώ τώρα εδώ εσείς συνεννοείστε και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω όμως διαπιστώσει ότι η κυρία Κάρλα Πέις έχει, ε, έχει εκδώσει ένα δεύτερο πρόγραμμα εργασίας, ενώ ο Μπράιαν ένα σχέδιο ε, λεπτομερές εφαρμογής. Και η διαφορά ποια είναι, το ίδιο πράγμα είναι. Έχετε πάρει διαφορετικό δρόμο ή είστε στην ίδια πορεία, οι κυρίες και οι κύριοι εκεί. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για την κυρία Πέις. Τι γίνεται τώρα με ε, την βυθοκόρηση του Δούναβη ε, στα TNT ημερίδες στο Ρότερνταμ. Ε, μάθαμε ότι αυτό είναι συντήρηση, αλλά όταν έχεις βυθοκόρηση στο Δούναβη είναι ολόκληρη επένδυση. Και ε, το έχουμε συζητήσει ε, με τους διαδρόμους TNT ότι οι επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται από το TNT, από το Connecting Europe Facility κτλ. Και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται εκεί και τι γίνεται με τη συνεργασία Ρουμανίας-Βουλγαρίας. Γιατί ο Δούναβης ε, είναι σύνορο των δύο χωρών και φαίνεται ότι δεν λάμπουν ε, δια της συνεργασίας τους οι δύο χώρες, για να το πω φιλικά. Ελπίζω η κυρία Πέις ε, να κάνει πρόοδο, έχει ήδη κάνει όπως βλέπω. Και τι γίνεται με τα χρήματα από τα Ταμεία Συνοχής. Αυτό είναι πάντα μία πρόκληση. Πώς συνδέονται αυτά. Μπορεί η κυρία Πέις τώρα ε, να χρησιμοποιήσει επαρκώς τα χρήματα από τη συνοχή. Ιδιαίτερα όταν ακούμε ότι υπάρχει υποαπορρόφηση. Τι γίνεται. Πιάνουν τόπο εκεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχω και τρεις ακόμα ερωτήσεις, αν μπορώ, προς τον κύριο Μπράιαν Σίμψον. Πρώτον, ποιες είναι οι συνέπειες της Συμφωνίας των Διεθνή Οργανισμών Ναυτιλίας σε σχέση με την, ε, το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Έχει συζητηθεί και έχει συμφωνηθεί στον IMO το 2023 να έχουν ε, και να καταθέσουν όλα τα στοιχεία για τις εκπομπές και τη ρήπανση. Αυτό θα έχει επιπτώσεις για σας κύριε Σίμψον. Δεύτερον, πριν από λίγες, λίγους μήνες, Πρόεδρε, συζητήσαμε την επικριτική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις επενδύσεις στους λιμένες. Και αυτή η έκθεση ήταν πραγματικά πολύ επικριτική και θέλω να ρωτήσω το Μπράιερ από τις τρεις επιλογές που μας παρουσίασε μήπως θα πρέπει να βάλουμε εκεί κάποιες προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες σε σχέση με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ξέρω ότι η έκθεση αυτή δεν αφορά τα προγράμματα TNT, τα διευρωπαϊκά, προηγείται χρονικά, αλλά έχει και επιπτώσεις γιατί τρέχουν ταυτόχρονα. Λοιπόν, και τρίτο, ε, αυτό που λέει ο Μπράιαν ε, στο σχέδιο λεπτομερές εφαρμογής, για τις θαλάσσιες λεωφόρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6% του γερμανικού στόλου ε, είναι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο ε, εκτός της Ένωσης. Λοιπόν, τι γίνεται με τις θαλάσσιες λεωφόρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι διάσταση αυτό ε, έχει, τι τάξη μεγέθους δηλαδή είναι αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ματενκάμπ. Κύριο Στέλιτσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω τους δύο προσκεκλημένους. Μετά από το δεύτερο αυτό γύρο παρουσιάσεων από συντονιστές μας, αν ε, έχω ένα, ε, μια εντύπωση, είναι ότι βλέπω να υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση ε, και συνεργασία μεταξύ των συντονιστών. Φαίνεται δηλαδή να δημιουργούνται κάποια κλάστερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ένα θετικό δείγμα. Ποιος είναι ο στόχος όμως αυτών των αλληλεπιδράσεων. Και εμείς καλό είναι που ενημερωνόμαστε για το τι γίνεται στα ευρωπαϊκά δίκτυα εν γέννη και στους διάφορους φακέλους που σας απασχολούν και τους διαδρόμους που εξετάζετε με αυτό το πλαίσιο, το πλαίσιο αυτής της αλληλεξάρτησης. Είναι σημαντικό να έχουμε την ανάλυση αυτή, το input επίσης σημαντικό. Γιατί μπορούμε και εμείς και από νομοθετής και από πολιτικής πλευράς να επηρεάσουμε κάποια θεωρητικά έγγραφα είτε ως ε, μεμονωμένοι βουλευτές είτε ως ομάδες βουλευτών. Είτε ω τα κράτη-μέλη που γνωρίζουμε καλύτερα. Θα ήταν καλό λοιπόν για όλους αυτούς τους σκοπούς και έχουμε λάβει δύο πολύ αναλυτικές παρουσιάσεις πληρέστατες, για να μην πω εξαντλητικές. Κάτι που λείπει όμως, δεν ξέρω μπορεί εγώ να μην το πρόσεξα, ποιο είναι το βασικό πολιτικό μήνυμα που θέλετε να μας περάσετε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το κατάλαβα, αλλά θα ήθελα να ακούσω τρία-τέσσερα βασικά συμπεράσματα που έχετε για μας. Και τελικά εμείς με ποιο τρόπο μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να ξεκαθαρίσω και στις συζητήσεις που θα έχω και στη συνέχεια. Μπορεί να μην πρόσεξα επαρκώς ε, τα λόγια σας, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το μήνυμά σας. Ένα input ε, πάνω στο οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Πριν τρία χρόνια ήμουν στην άλλη πλευρά, τώρα είμαι εδώ, ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι το έργο των συντονιστών και οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε ενίοτε. Βλέπω πάντως καλύτερη εστίαση, συγκέντρωση και αλληλεπίδραση από ό,τι μέχρι τώρα και ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τέλιτσκα, ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ για τις δύο παρουσιάσεις η ε, εσωτερική ναυσιπλοεία και η ναυσιπλοεία ε, ανοιχτής θαλάσσης δεν είναι πάρα πολύ φιλική στο περιβάλλον. Και η λύση είναι να προσαρμοστούν τα σκάφη προς τους ποταμούς και όχι το αντίθετο, το, αντίθετο, ε, το αντίστροφο και στη θάλασσα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις εκπομπές. Ε, ο σιδηροδρομός που είναι φιλικός προς το περιβάλλον πληρώνει διάφορα τέλη ενώ η ε, ε, ναυσιπλοεία εξαιρείται. 80% της εσωτερικής ναυσιπλοείας στην Ευρώπη είναι στο Ρήνο αλλά 80% των χρημάτων πηγαίνουν αλλού στη Γερμανία ξέρω τι φταίει. Έχουμε τρεις ε, διοικήσεις ε, για κάθε θέμα της εσωτερικής ναυσιπλοείας που κάθε μια φτιάχνει τρία προγράμματα. Σύλλογο 9. Παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια στη Γερμανία ε, αποφάσισε ότι χρειάζεται ένα νέο λιμάνι. Γιατί ο Έλβας δεν είναι αρκετά βαθύς και προς τη Βέζα για να μην πηγαίνουν όλα στο Ρότερνταμ να πηγαίνουν και στο Αμβούργο. Δύο μεγάλα πλοία έφτασαν και τώρα πρέπει να βυθοκορηθεί και να σκάψουν τον Έλβα. Εχθές διάβασα ένα άρθρο στην εφημερίδα που λέει ότι φοβάται το λιμάνι του Βίλεμς Χάφεν ότι όλα θα πάνε στο Αμβούργο και ότι θα πάει στο Βρόντο όλο το λιμάνι, θα μείνει αχρίαστο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι τρελά πράγματα. Είτε θα φτιάξουμε νέο λιμάνι, είτε θα σκάψουμε να βγάλουμε να βαθύνουμε τον Έλβα και τα δύο είναι ε, σπατάλι και ήρθε το εδώ ελεκτικό συνέδριο και μας τάψαλε και είπε ότι έψαξε ε, όλα τα προγράμματα και τίποτα δεν έβγαλε αυτό που είχε ε, προβλεφθεί. Δηλαδή είναι οικονομική καταστροφή. Λεφτά έχουμε αρκετά, αλλά το θέμα είναι πώς τα επενδύουμε. Αν τα επενδύουμε σωστά. Άλλο παράδειγμα. Φυσικά, πολύ ωραίες οι συνδυασμένες μεταφορές και Brian θα θυμάστε στα TNT δίκτυα στο παρελθόν τα διευρωπαϊκά είχαμε πει θέλουμε σύνδεση 40 ε, ε, χιλιόμετρα στη Νίκαια ε, να φτιάξουμε ένα κομμάτι που λείπει για να φτάσει μέχρι την Κοπεχάγη που είναι ο πιο σύντομος δρόμος να πηγαίνει με το τρένο το εμπόρευμα από τη Μεσόγειο στην Κοπεχάγη. Ε, αντιστάθηκε η ιδανική κυβέρνηση γιατί θέλει να προωθήσει τα λιμάνια της. Και αυτά είναι τρελά τα πράγματα. Πάμε στην αυσιπλοεία, ενώ η ναυτιλία δεν είναι φιλική προ το ε, περιβάλλον και αφήνουμε το σιδηρόδρομο. Θέλουμε να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα την ναυτιλία, να τη δώσουμε ευκαιρία. Αναφέρθηκε και στι εκπομπέ. Και παίζει ρόλο και η μεθανόλη και το ε, ε, υγραέριο. Χωρίς τεχνική καινοτομία θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαιρετικά φιλική στο περιβάλλον την εσωτερική να ψηπλώει. Εγώ δεν είμαι φίλος του Diesel, πόσο μάλλον μετά το Gate. Αλλά αν θέλουμε να φτάσουμε στο μισό της εκατό από το 2020 για το ε, αργό πετρέλαιο, το βαρύ πετρέλαιο, έχουμε ακόμα 500 φορές περισσότερους ρήπους από ότι στο ντίζελ. Μπορούμε να απαγορεύσουμε ε, το βαρύ πετρέλαιο που έτσι είναι ένα κατάλοιπο, ένα απόβλητο των δηληστηρίων ε, για να ε, βελτιώσουμε σημαντικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και να περιορίσουμε τους ρήπους. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, αναβάλουμε 2020 κτλ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το υγραέριο. Μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, αλλά το σημαντικό είναι να σταματήσουμε το βάρη πέτρα αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, ακόμα και αν περάσει το μισό της εκατό, δεν ξέρουμε πώς θα το ελέγχουμε. Έτσι κι αλλιώς ε, περιμένουν ε, τα πλοία να βγουν 10 χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι και μετά αρχίζουν τις εκπομπές. Πολύ θετικό παράδειγμα επίση στην Ευρώπη δεν έχουμε μόνο στρατηγική για τη Βαλτική αλλά και τη στρατηγική για το Δούναβι. Και οι χώρες που βρέχονται ο δούναβη, που είναι 10 δεν είναι μόνο οι άμεσε, θέλουν να συνεργαστούν, όχι να φέρνουμε αντιμέτωπα λιμάνι με λιμάνι, κράτος με κράτος ε, θέλουν την προοπτική να συνεργαστούν προ την κατεύθυνση αυτή. Και το λένε. Έχουμε παραδείγματα Είχε πάει ε, στα πέντε λιμάνια από τρία κράτη που συνεργάζονται γιατί δεν θέλουν να έχουν ανταγωνισμό αλλά συνεργασία. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση να πάμε. Αλλά δεν καταφέρουμε αυτό να κάνουμε στη Γερμανία. Φαντάσου στην Ευρώπη. Χαίρομαι πιο πολύ για τη στρατηγική του Δουνάβιος γιατί μας δείχνουν το δρόμο και θα μπορούσε η Ευρώπη να μάθει πάρα πολλά. Η Γερμανία, συγγνώμη, από την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητής. Τέλει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι. Σειρά μου δεν ήταν. Γιατί κοιτάτε αλλού. ναι, εσείς είστε. Η σειρά σας είναι. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ καλά, πολύ που βλέπω τους συντονιστές Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση, ιδίω για τον Δουναβή. Είμαι Ούγκρος, δεν έχουμε δυστυχώς θάλασσα εμείς, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό με ενδιαφέρει ο Δούναβης πιο πολύ. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που αναφέρατε τις περιβαλλοντικές πτυχές. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η βιοπικιλότητα, η διατήρηση των εθνικών οικοσυστημάτων είναι προτεραιότητα για τα παραδονάβια κράτη, όπως το δικό μου. Αναφερθήκατε στη Σερβία αρκετές φορές ε, στην παρουσίασή σας. Γιατί γίνεται λόγος για αυτό το διδικτυακό αποτέλεσμα και φυσικά και πρέπει και η Σερβία να συνεργάζεται για αυτό το διάδρομο. Στην παρουσίασή σας μας δείξατε εικόνες ε, για κάποια συστήματα, ε, για κάποια πλοία, ψηφιοποίηση. Όλα αυτά ενδιαφέρουσα τεχνολογία είναι και μπορούν να βελτιώσουν ε, την μεταφορά και την αυσπλοεία στο Δούναβι. Δεν θέλω να επανέλθω. Υπάρχει κάποια διασύνδεση όμως, γιατί μιλήσατε για τη Βαλτική σε σχέση με την Κροατία και είπατε κάτι για τη Βουλγαρία. Μετά δεν ξέρω, υπάρχει κάτι στο μέλλον στο μεταξύ. Στην παρουσίασή σας επίσης ε, αναφερθήκατε στη συνάντηση των Υπουργών ε, Μεταφορών στο Ρότερνταμ. Κατά την δική σας άποψη, τι είναι το πιο επίγον, ποια είναι η πιο επίγουσα προτεραιότητα για το μέλλον των ευρωπαϊκών δικτύων στον των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά το Δούναβι συγκεκριμένα. Τι πρέπει να συμφωνήσουν οι Υπουργοί Μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέλη. Εσείς. Thank you, Madam Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσω τους διαμιλητές ε, και να τους ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις τους. Ιδίως για τις θαλάσσιες λοφός αυτά που είπε ο Μπράνι Σίμψον, μας ε, ε, μιλήσατε για τους τρεις τομείς οποίους θα εστιάσετε. Και επίσης η αλυσίδα της εφοδιαστικής και οι θαλάσσιες μεταφορές στην παγκόσμια αλυσίδα, κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για τα περιφερειακά κράτη και ότι καλό είναι να συνδέσουν τις προσπάθειές τους και να μην κάνει το καθένα τα δικά του για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τους φραγμούς ε, και να μπορεί να υπάρχει ελεύθερο εμπόριο. Ιδίως στο πλαίσιο του Brexit τώρα, εγώ είμαι από την Ιρλανδία και αντίθετα από ό,τι είπε ο προλαλής σας, εμείς μόνο από θάλασσα βρεχόμαστε και επομένω μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε τους ε, φραγμούς και τα κενά που υπάρχουν είπατε θα εστιάσει τον περιφερειακό χαρακτήρα συγκεκριμένα. Θα δώσετε περισσότερη έμφαση λοιπόν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίω εν ώψη του Brexit, γιατί κάποιε χώρε θα θυγούν και καλό θα ήταν να υπάρξει επιπλέον υποστήριξη περιοχή αυτές για να γεφυρωθούν ε, τα προβλήματα και τα κενά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε τι παρουσιάσεις. Δεν είμαι βέβαια και τόσο αισιόδοξη, αλλά τέλος πάντων. Το χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030 είναι μια τεράστια πρόκληση. Εγώ έρχομαι από την Αυστρία και βλέπω στη χώρα μου ότι φυσικά και έχουμε προβλήματα για τον Δούναβη, για το πολυτροπικό τερματικό που δεν υπάρχει σε εμά και μάλλον δεν θα έχουμε και σύντομα. Έχουμε για, το, για τα τρένα ένα εμπορευματικό σταθμό, αλλά έχουμε προβλήματα και με τις γειτονικέ χώρες και στην Επιτροπή μας το έχουμε συζητήσει με το ERTMS και τον ανταγωνισμό που δεν βλέπουμε να λειτουργεί ομαλά στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ε, εξακολουθεί να επικρατεί ε, το, η τάση της κρατικοποίησης των σιδηροδρόμων. Σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση που αναφέρατε, Εμεί ε, στην Αυστρία έχουμε το Ομοσπονδιακό Σιδηρόδρομο και έχουμε προσπαθήσει ένα μεγάλο τμήμα να εξυγχρονιστεί, ιδίω στα δυτικά και έχουμε και κάποιες δοκιμαστικές ε, τροχίες και για αυτοκινούμενα οχήματα. Ε, υπάρχει μεγάλη ε, που δίνεται στο οδικό δίκτυο ε, σε αντίθεση με τους σιδηροδρόμους και αυτό είναι κάτι κατάφορο. Το θέμα είναι εσείς πώς θέλετε να το αντιμετωπίσετε και να το αναστρέψετε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή πώς ε, θα προσπαθήσετε να επηρεάσετε και τα κράτη ώστε να υπάρξει διασυνοριακή πολυτροπικότητα και σχετικά δίκτυα. Merci beaucoup, Madame Schmidt. Alors... Ευχαριστώ. Κάρλα Μπράιαν. Πολλά ερωτήματα, αλλά επαναλαμβανόμενα. Πώς θα εργαστείτε με τα κράτη-μέλη. Ήταν κάτι που το είπε και ο εισηγητής, ο κύριος Ισμαήλ Ερτούκ, που είπε ότι ναι, υπάρχουν και επιτόπου κάποια project που τα επισκεφθήκαμε. Είδαμε συγκεκριμένα αυτό το project για τα φρούτα που έρχονται από το Ισραήλ στη Μασαλία. υπήρξαν και πραγματικά ερωτήματα, να φέρθηκε το Brexit και τι γίνεται και με τις θαλάσσιες αυτές αρτηρίες ε, και με τα, ταμείο, με τα ταμεία συνοχής, τα κονδύλια του ταμείου συνοχής. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και η διασύνδεση μεταξύ των προτεραιοτήτων και το τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο στην έκθεσή του, που δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Το πολιτικό μήνυμα ποιο είναι, το συμπέρασμα ποιο είναι, που, τι πρέπει να συγκρατήσουμε. Ακούσαμε και τον κύριο Κράμερ πόσο σημαντικό είναι το θέμα των εκπομπών. Τι θα κάνετε με το σχέδιο δράση και με τη στρατηγική για τον Δούνα. Ο κύριος Ντέλη μίλησε για τη βιοπικιλότητα και τους οικοτόπους και ζήτησα να μας πείτε στην διάσκεψη αυτή κορυφής ε, ιδίως το διάδρομο του Δούναβη, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα προωθήσετε. Σας είπε η επόμενη συνάδελφος, μην ξεχνάτε τις περιφέρειες. Γιατί με τον Brexit, ιδίω τώρα είναι που δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε. Επίσης είπε η κυρία Σμίτ ότι είναι μεγάλος ανταγωνισμός ε, του συνδρομικό δίκτυο στην Αυστρία, ε, όπου μεγαλύτερη βάρτια δίνεται τις οδικές μεταφορές και κατά πόσο θεωρείται ιδιαίτερα αισιόδοξη την προθεσμία του 2030. Φτάνουν αυτά ή θέλετε κι άλλα. Ποιος θα ξεκινήσει, Επτά λεπτό καθένας περίπου έχετε. Επτάμιση, λέει η κυρία Πέις. Εντάξει, επτάμιση. Λοιπόν, Κάρλα, ξεκινάτε εσεί. Ε, το κύριο Ερτούκ. Και ο κύριο Βαντενκάμπ. Μιλήσατε για το Brexit και το Ενώμενο Βασίλειο. Έχουμε την πολιτική μας, αλλά δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Σχέδιο δράσης και λεπτομεριακή εφαρμογή. είναι ακριβώ το ίδιο. Απλά έχει διαφορετικό όνομα Ουσιαστικά περί του ίδιου πράγματο πρόκειται. Σχέδιο υλοποίηση, σχέδιο δράση, ε, τα ίδια είναι ουσιαστικά. Γιατί ο στόχο είναι να αντιλοποιήσουμε και τα δύο στο τέλο για τη βιδοκόρηση του Δούναβη. Ε, συνεχίζεται η διαδικασία αυτή. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Και η συντήρηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, γιατί τη βυθοκόρηση δεν χρηματοδοτούμε. Αυτό που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όμως είναι τα πλοία. Αν έχω βιδοκορήσει το την Κίτη. Ε, έχω μετά ένα ε, μηχάνημα μέτρησης που σε πραγματικό χρόνο μετρά μπορούμε να φέρουμε ειδικά σκάφη να μετρήσουμε τους τόνους που μπορεί να περνάνε κτλ. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Έχουμε κονδύλια από τη γάμα δέλτα μουβ και από τη γάμα δέλτα ρέγγιο. Ε, Άρα ουσιαστικά όταν λέμε για βυθοκόρηση μιλάμε για συντήρηση. Είναι σαν να πηγαίνει στο τζαγκάρι με τα παπούτσια σου και θέλεις, ε, ε έχεις αγοράσει καινούργια και πληρώνεις δάνειο για τα παλιά ακόμα. Κάτι τέτοιο. συνεργασία μεταξύ Ρουμανίας Βουλγαρίας. Πράγματι. Κάποια χρόνια της ζωής μου τα δαπάνησα για να κάτσουν στο δύο τραπέζι κάποιες χώρες μεταξύ τους να τα βρουν. Το Φεβρουάριο συνάντησα τους δύο νέους υπουργούς. Και Ο Βουλγαρος Υπουργός έκανε ένα θαύμα. Είχε έναν τριετή προπολογισμό για τη βυθοκόρηση, είχε αυτό το σκάφος μέτρησης, προκήρυξε διαγωνισμό και αγοράζει και ένα σκάφος βυθοκόρησης. Τρία χρόνια. Μήνα μάφωνη. για το τι πέτυχαν στα τρία χρόνια. Οι Ρουμάνοι διαφορετικό. Επειδή έχουν πάρα πολλέ καταγγελίε από του παικτέ και τα λοιπά, έχουν πρόβλημα με τη βυθοκόρηση κάθε χρόνο. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί βέβαια, γιατί τώρα έχει αλλάξει ο υπουργό. Έγιναν πριν δύο εβδομάδε εκλογέ στη Βουλγαρία ε, και ελπίζω φέτο να ξεκινήσει βεθοκόρηση πριν το καλοκαίρι και θα είναι κάτι καταπληκτικό. Έτσι πιστεύω. Και ελπίζω να βγω και αληθινή. Ταμείο Συνοχής, όταν ξεκινήσαμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, είχαμε 11,1, 11,3 δις από τη γαμαδελταρέγγιο για ε, από τις χώρες περιφέρειας και αυτά έχουν σχεδόν δαπανηθεί εξ ολοκλήρου. Ή τέλος πάντων όχι δαπανηθεί αλλά διατεθεί για τα διάφορα project. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στις χώρες συνοχής για όλα τα project και για τα κονδύλια αυτά. Γιατί τώρα τα έχουμε, αλλά του χρόνου δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άρα τώρα που υπάρχουν θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Έτσι σκέφτονται τα κράτη. Άλλο γενικό προβλήματος, άλλο τα κονδύλα συνοχή. Πάβελ. Είπες ποια είναι τα βασικά project. Θα έλεγα το εξής. Τουλάχιστον διτροπικότητα για να μην πω πολυτροπικότητα διασυνοριακό επίπεδο μας ενδιαφέρει πολύ. Γιατί βλέπω ότι κάθε χώρα, όπως και δική μου, επικεντρώνεται στα δικά της. Δηλαδή ασχολείται με τους επιβάτες στη δική της χώρα. Έχουμε όμως και το διασυνορικό επίπεδο και υπάρχουν ε, οι διαφορές. Μπορεί να είναι διαφορετικοί οι κανονισμοί, τα ψηφιακά συστήματα μεταξύ των όμορων ε, χωρών, να υπάρχει ένα πρόβλημα με τη γλώσσα κτλ. κτλ. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι η βιωσιμότητα. Πώς θα είμαστε βιώσιμοι. Χρειαζόμαστε καλύτερα κάψιμα, χρειαζόμαστε ψηφιοποίηση. Θέλουμε ε, ανακαίνιση των κτηρίων, θέλουμε ειδικό σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να είμαστε παντού. Πρέπει να κάνουμε κλάστερ και σχέδια. Αυτά νομίζω είναι τα σημαντικότερα για τα διευρωπαϊκά Συντομέτα μεταφορών αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι για τα τρένα KPI. Τα KPI είναι τα ίδια τα συστήματα ασφαλείας δεν είναι τα ίδια. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά. Για τον κύριο Κράμερ. Πόσο χαίρομαι. Τέταρτη φορά, τη πω πέμπτη, μάλλον πέμπτη χρονιά, έρχομαι και είναι η πρώτη φορά που μιλήσετε για την εσωτερική ναυσιπλοεία. Και είπατε ότι είναι φιλοπεριβαλλοντικός αυτός ο τρόπος μεταφοράς. Θα σας φιλήσω. Θα σας φιλήσω μετά. Μετά, όχι τώρα. Okay. <laughs> Μετά, έτσι. Μετά, λέει κύριε Αντελή, όχι τώρα. Μπορείτε να μου κάνετε όμως μια χάρη. Να ζητήσετε από τη Γερμανία να αναστείλουν την, ε, το μπλοκάρισμα. που μας δυσκολεύει με το Δούναβι. Αν θέλουμε να περάσουμε σε καθαρά πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα με το βαρύ πετρέλαιο. Μην το ξεχνάτε. Υπάρχουν κάποια δηληστήρια που εξεργάζονται το βαρύ πετρέλαιο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πού το βάζεις. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας στο βαρύ πετρέλαιο, να το προσέχουμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για το βαρύ πετρέλαιο. Για να μην μολύνει το περιβάλλον, να μην εκτεθεί στο περιβάλλον. Και είναι και τεράστιες ποσότητες. Άρα πρόκειται για μια μεγάλη περιβαλλοντική πρόκληση. Για τον κύριο Ντέλη. Ναι, το περιβάλλον πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να σας πω τι κάναμε πρόσφατα, τον τελευταίο χρόνο. Είχαμε ένα δεν πυρογνωμόνων. Αν μια χώρα έχει ε, δυσκολίες με ένα project και θέλει κατάρτιση για το προσωπικό της, για να μπορεί να δει τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σε σχέση και με την εθνική, μπορεί να ζητήσει βοήθεια από αυτήν την ομάδα πυρογνωμών. Και μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι πιστεύουμε τουλάχιστον για να διευκολυνθεί πολύ όλη η διαδικασία. Όλες οι χώρες και οι χώρες συνοχής έχουν έλλειψη προσωπικού που να ξέρουν καλά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που είναι και πολύ το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι και από τις χώρες μας ο καθένας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, υπάρχει λοιπόν αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων. Και όποιος τους θέλει μπορεί να ζητήσει τη βοήθειά τους. γιατί έχουμε τον καλονισμό, τον περιβαλλοντικό και για τον Έλβα και πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Τι κάνουμε τώρα. Κατεπηγόντω, αυτό ρωτήσατε. Ποιο είναι το πιο κατεπήγον για μα αυτή τη στιγμή. Νομίζω την απάντηση την έδωσα απαντώντα τον Πάβελ. Περιβάλλον, νομοθεσία, διασυνοριακό επίπεδο. Αυτά τα θέματα που ανέφερα πατώντας στον Πάβελ. Ιρλανδία. Που είναι απομονωμένη και πρέπει να φτιάξουμε γέφυρες. Ναι, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια γέφυρα. Για την κυρία Σμιτ. Με το βήμα και πράγματα Έχουμε πρόβλημα Ο Δούνευς είναι ένας πολύ ζωντανός ποταμός, πολύ όμορφος ποταμός. Το πρόβλημα είναι πώς θα παραμείνει έτσι, να μην κάνουμε μεγάλη παρέμβαση όμως ταυτόχρονα. Και με τη βυθοκόρηση να μην το παρακάνουμε, για να μπορούμε να τον επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση μετά. Είπατε ότι είσαι από την Αυστρία. Καλά, δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι τα πήγε πολύ καλά η Αυστρία. Και το λιμάνι της, Φιένα, της Βιέννης πάρα πολύ καλά πηγαίνει. Αλλά για τη βιβλιοκόπηση πράγματι υπάρχει ζήτημα. πρέπει να δούμε. Οι εργασίε βιδοκόρηση αν είναι νόμιμε, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε κάτι παράνομο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για όλε τι απαντήσει και τώρα ο λόγος στον κύριο Σίμψον. Ευχαριστώ. Ισμαήλ. Ήμουν 25 χρόνια στο Κοινοβούλιο και το πρόβλημα ήταν επί 25 χρόνια τα κάτι μελη Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να τους χτυπάμε διαρκώς με το σφυράκι αυτό της υπομονής. Σίγουρα κάποια χώρα θα έχει μια προτεραιότητα που δεν την έχει και διπλανή, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε, να πιέσουμε για να συμμετάσχουν στο όλο εγχείρημα. Το όλο εγχειρήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, συνολικά, όχι μόνο οι θαλάσσιες λεωφόροι ή οι διάδρομοι ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά Συνήθω τα κοιτάνε τα κράτη-μέλη από τη σκοπιά τη δική του, αν περνάνε τι χώρε του. Εμεί όμω είμαστε οριζόντιοι και όχι κάθετοι. Αυτή είναι και η δυσκολία. Αυτή είναι η προσέγγιση μα. Οπότε το γνωρίζω Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε πιστικοί και να ε, πάρουμε, να συμπαρασύρουμε τα κράτη-μέλη στην όλη μας προσπάθεια. Για τον διάδρομο που ανέφερα στην ομιλία μου, για τον ε, διάδρομο της ε, φρέσκιας τροφής, για τα προκυπευτικά ε, κάποια φορτία ε, φρούτα πηγαίνουν προς τη μία κατεύθυνση και τα άλλα πάνε προς την άλλη, ώστε να είναι κερδοφόρα η όλη ε, διαδικασία για, τα, για τους σιδηροδρόμους. Και με τους απαραίτητους διάβλους. Πάρτε κοιτάμε και στο Ισραήλ και στην Ιορδανία είναι απλώς ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ως τώρα πάει καλά. Ε, πάντως, να σας, ε, θα σας κάνω, θα σας εκπλήξω ίσως, να σας πω ότι εμείς θα θέλαμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εδώ έχουμε μια αποσύνδεση όπως είπε και ο κύριος Κάλλας, ε, ε, η Βρετανία θα είναι μια γειτονική χώρα, σαν το Μαρόκο. Η Νορβηγία τα πηγαίνει καλύτερα. Θα υπάρχει ένα πρόβλημα με την Ιρλανδία βέβαια, αλλά αυτό το σχολιάσω αργότερα. Η έκθεση του Ολυμπικού συνεδρίου δεν μιλούσε μόνο για τις προμήθειες στα διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά γενικότερα για το θέμα των προμηθειών. Εφόσον το ΣΕΦ άρχισε να λειτουργεί, η διευκόλυνση για τη διασύνδεση της Ευρώπης, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και κοιτάζουμε τις επενδύσεις ε, με περισσότερο ορίζοντα το μέλλον. Νομίζω πάντως ότι το ελεκτικό συνέδριο ήταν λίγο εκτός θέματος όταν μας επικρίνανε. Το ίδιο και με το ERTMS. Κοιτάζουν λίγο το τελικό αποτέλεσμα απλώς στο ελεκτικό συνέδριο καμιά φορά και ε, εκτό από τον τελικό λογαριασμό υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες. Κύριε Τελίτσκα, για τους διαδρόμους. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, συνεργαζόμαστε. Και έχουμε φάει νερό και αλάτι. Εδώ λοιπόν πρέπει να τονίσουμε τρεις πολιτικές προτεραιότητες. Περιβάλλον, θαλασσια θέματα και εφοδιαστική και ασφάλεια στη θάλασσα. Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες και δεν απομακρυνόμαστε ποτέ από αυτές τις τρεις πολιτικές προτεραιότητες. Μάικλ. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, διότι τα λιμάνια είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Οπότε, ε, οι μένες δεν θέλουν να ξέρουν τι κάνουν οι δε, ιδίως αν είναι κοντινά. Το Βίλεγξχαμ και το Αμβούργο λόγου χάρη, το Άμστερνταμ, το Λίβερπουλ και το Σαουθάμπτον, έχουν μια τέτοια στάση. Συμφωνώ. Δεν αξίζει να χτίσουμε ένα φοβερό λιμάνι στο Σορθάμπτον. Στο Βίλεμς Χάφεν ε, και να γίνει κάτι τελείως άσχετο κάπου κοντά. Ο καθένας κοιτάζει λίγο τις δικές του ανάγκες εγωιστικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, σημειώνω πάντως αυτό που είπατε και αυτό έχω εγώ να σχολιάσω. Βιμ, Μάικλ, μάλλον. Τα θαύματα θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο. Θέλουν το χρόνο τους. Κοιτάζουμε πώς θα υλοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο την οδηγία του ΑΕΜΟ. Και θα τεθεί σε ισχύ λογικά το 2020 παρόλο που υπάρχει ένα ερωτηματικό για το τι θα γίνει με τους σταθμούς υγροποιημένου αερίου, ε, πώς θα διευθυντήσουμε το θέμα της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας ως τότε. Όμως η δουλειά μας συνεχίζεται με το πρόγραμμα πρόληψης της ρήπανσης από τη σκοπιά του ΑΕΜΟ. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι για την υλοποίηση το 2020. και προσπαθούμε να προλάβουμε στο 2020, και το 2025, γιατί θα σημαίνει ότι έχουμε καθυστερήσει σε πολλά. Για τις περιφερειακές περιοχές έχουμε πολλά στοιχεία για τις ε, περιφερειακές περιοχές και μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποια έργα με ωφέλη κυρίως περιβαλλοντικά. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Για τις περιφερειακές περιοχές συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα όπως TRDF και τα προγράμματα συνοχή. Εκεί δίνεται έτσι κι αλλιώ ιδιαίτερη προσοχή στι περιφερειακέ περιοχέ. Πάντως, στα πλαίσια της δικής μας ε, ε, εντολής και αρμοδιότητας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αναγκαστικά δεν μπορούμε να δώσουμε όλη την ε, δέουσα προσοχή στις περιφερειακές περιοχές, γιατί μας ενδιαφέρει τι γίνεται διασυνοριακά και το καθεξής. Βέβαια, ε, έχω υπόψη μου ότι οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και θα το συζητήσουμε ίσως πληρέστερα όταν περάσουμε στην φάση της αξιολόγησης και συζητήσουμε τις ανάγκες ακριβώς των περιοχών της περιφέρειας. Δεν το απορρίπτουμε λοιπόν, απλώς δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Κυρία Κλούν, όντω πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της Ιρλανδίας. Όμω όταν φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα γίνει ακριβώ. Θα είναι πολύ δύσκολο. Υπογραμμίζω όμω αυτό που είπα και τώρα για την περιφερειακή διάσταση. Θα λάβει τελείω νέο νόημα η περιφερειακή διάσταση με αυτή τη μεγάλη τρύπα που θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο στο χάρτη τη Ευρώπη. Και ναι, και η Βόρεια Ιρλανδία θα είναι μια σκιά και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να το δούμε αργότερα και να βρούμε έναν τρόπο η Ιρλανδία να αισθάνεται διασυνδεδεμένη με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό και γι' αυτό ασχολούμαστε και με τις περιφερειακές περιοχές. Δεν είναι μόνο οι Αζόρες και τα μακρινά νησιά, οι απόκεντρες περιοχές, οι περιφερειακές, είναι και άλλα πράγματα. Και σε δύο χρόνια μπορεί να γίνει και η Ιρλανδία περιφέρεια της Ευρώπης. Κύριε Σμιτ, κυρία Σμιτ, είπατε να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι. Ε, ούτε για το διάδρομο του Δούναβη, ούτε για την πολιτική των ευρωπαϊκών δικτύων. Εγώ είμαι απλώ αισιόδοξο. Δεν είμαι ούτε μη αισιόδοξο ούτε κάτι άλλο. Για πρώτη φορά έχουμε μια πολιτική συνεκτική για τα ευρωπαϊκά δίκτυα σε όλη την Ευρώπη που μπορεί να δώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν είμαι λοιπόν υπεραισιόδοξο ε, για τα θέματα γενικότερα που αναφέρατε, αλλά είμαι συγκεκριμένα αισιόδοξο για το θέμα αυτό. Ναι, υπάρχουν λιμάνια που δεν θέλουν να πάρουν μέρος στη συνεργασία μας. Κοιτάζουν να κάνουν μόνο τη δουλειά τους. Όμως, εάν μιλάμε για Ευρώπη, είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να ακολουθήσουμε την πολιτική των ευρωπαϊκών δικτύων. Μπράιαν, Κάρλα, σας ευχαριστούμε που παραμένετε αισιόδοξοι. Πάντως, η Επιτροπή Μεταφορών είναι στο πλευρό σας, παραστάτης. Θα παρακολουθούμε και τα θέματα του Δούναβη και της θαλάσσης Λεωφόρους και την εξέλιξή σου. Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις των καθένα μας ξεχωριστά και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι ε, στην Επιτροπή σας και θα σας υποστηρίξει το Κοινοβούλιο. Θα παρακολουθεί πολύ στενά τις εργασίες. Ε, συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας και στο επανειδήν.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 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ένα θέμα συναρπαστικό που μας θυμίζει τα νιάτα μας όλους και τα παιδικά μας χρόνια. Στρατηγική διαστημική για την Ευρώπη. Θα δώσω μέσα στο λόγο Η συγκήτριά μας, η κυρία Μάισνερ, δυστυχώς κολλείεται και αποσιάζει. Περιμένουμε να κάνει ε, ο κύριο Σίμψον εδώ τη βόλτα του να χαιρετήσει διαφόρου Γεια σα. καλημέρα σα, Ε, τι να κάνουμε, πρώην πρόεδρος επιτροπή Μεταφορών είναι. Τι να του πω, εγώ το σέβομαι και είναι και φίλο μου. Voilà, Να τελειώσουν οι αναγκαλισμοί και τα φιλιά. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εγώ ήθελα να βάλουμε λίγη πίεση εδώ στην Επιτροπή μας μιλώντας για το διάστημα και ε, θυμηθούμε και τα παιδικά μας χρόνια, αλλά μάλλον απέτυχα ικτρά. Λοιπόν, η κυρία Μάισνερ δυστυχώς η συγγήτρια ε, κολλείεται και αποσιάζει. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τέλιτσκα για να μας παρουσιάσει την έκθεση της κυρίας Μάισνερ για τη διαστημική στρατηγική της Ευρώπης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, θα σας παρουσιάσω κάποια σημεία που θα σας έλεγε η Γκεζίνε Μάισνερ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε γιατί είχε μια άλλη ανελημμένη υποχρέωση. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι μια τέτοια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της διαστημικής ε, στρατηγικής είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό λέει και η συγκήτριά μας. Η Ευρώπη έχει παγκοσμίω ένα μερίδιο 21% πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή ε, των ετησίων κερδών και 230.000 εργαζομένους στο διαστημική βιομηχανία. Δηλαδή είναι από τους παγκόσμιους ηγέτες. Αλλά πόσες φορές το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, το έχουμε ξαναδεί σε διάφορους κλάδους που ήμασταν ηγέτες και τη χάσαμε αυτή την πρώτο καθεδρία μας. Οπότε να μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Οι διαστημικές τεχνολογίες ε, είναι επίσης ένα άλλο στοιχείο που παίζουν ε, παίζει σημαντικό ρόλο και θα εξακολουθεί να το πράττει και στο μέλλον. Γι' αυτό ο ε, στόχος της νομοδότησης είναι να τονίσουμε ε, το ρόλο των μεταφορών στη στρατηγική αυτή για το διάστημα. Έρχομαι τώρα στην ουσία της νομοδότησης. Μερικά σημεία επιγραμματικά να μοιραστώ μαζί σας. Η γνωμοδότηση τονίζει την προσέγγιση φιλική προς την τεχνολογία, ότι οι μεταφορές θα πρέπει να είναι τμήμα των μελλοντικών αποφάσεων για το διάστημα. Γι' αυτό η Γκεζίνε Μάισνερ ενθαρρύνει τους ενδιαφερομένους των μεταφορών να συμμετέχουν στο διάλογο με τον κλάδο της διαστημικής βιομηχανίας και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό και θέλω να το υπογραμμίσω κι εγώ. η αλληλοδίζηση των διαφόρων κλάδων της ε, βιομηχανίας είναι κάτι που δεν έχουμε πάντα αρκετά στο μυαλό μας. Στη συνέχεια η γνωμοδότηση αναφέρει που μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις η διαστημική τεχνολογία. Λέει η κυρία Μάισνερ για τις συνδυασμένες μεταφορές, για την ανάπτυξη ε, των μεταφορών και των διαφόρων συστημάτων που έχουν ε, ε, μεγάλες προκλήσεις ε, για τα διαδίκτυα και τις συνδυασμένες μεταφορές, πολυτροπικές. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία. Η τεχνολογία που συνδέεται με το διάστημα θα παίξει ε, πρωταγωνιστικό ρόλο για τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους επιβάτες και θα βελτιώσει την υποδομή διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας με εναλλακτικά συστήματα ελέγχου και επικοινωνίας και τεχνολογίες για ε, αυτόματη απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών. Άλλο θέμα που αναφέρει η γνωμοδότηση. Πώς θα μεταφερθεί στο μέλλον, θα μεταφραστεί μάλλον η στρατηγική αυτή και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ο Επίτροπος Σεύσκοβιτς είπε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται θα αποδώσει επταπλάσιο ποσό. Ελπίζω να πω εγώ, αλλά αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το δυναμικό που υπάρχει. Η Γκεζίνε λέει ότι παραμένει να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κάνω και τα δικά μου σχόλια και δεν το έχω διαβάσει και βλέπω στην επόμενη σειρά ότι λέει ακριβώ τα ίδια η Γκεζίνε Μάισνερ. Βλέπετε φιλελεύθεροι πόσο ενωμένοι είμαστε και συνεκτικοί στις απόψεις μας. Ε, τα προϊόντα επίσης που έχουν να κάνουν και υπηρεσίε με την ε, ασφάλεια των μεταφορών, data streaming, ε, διαχείριση της κυκλοφορίας, ε, ένα ευέλικτο πλαίσιο εφοδιαστικής κτλ. Τρία ακόμα σχόλια πριν σταματήσω και προχωρήσω σε κάποια συμπεράσματα. Δίνεται ιδιαίτερη εστίαση στη γνωμοδότηση και προσοχή στην αυξανόμενη εξάρτηση των μεταφορών από τη διαστημική τεχνολογία όταν πρόκειται για την ε, διαχείριση ε, της κυκλοφορίας ή συστήματα εντοπισμού ε, των μεταφορών θα πρέπει να μεταφερθεί φυσικά και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ε, για την ε, μεταβίβαση δεδομένων, πάντα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και στην ιδιωτική ζωή. Και θα πρέπει να δούμε επίσης ε, τι γίνεται με το Γαλλία Ελαίο, που είναι στην τελική φάση της πλήρους ανάπτυξης, χρειάζεται ακόμα υποστήριξη για να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του, το δυναμικό, να υπάρχουν καινοτόμα πλαίσια. Όσοι είχαμε πάει στην αποστολή ε, πέρυσι για το Γαλιλαίο ξέρουμε τι εννοεί είναι. Είναι τεράστιο πραγματικά το δυναμικό και παραμένει ανεκμετάλλευτο σε μεγάλο βαθμό. Συμπεράσματα. Γενικά, ο κλάδος του διαστήματος είναι σημαντικός όχι μόνο για μεγάλες εταιρείες αλλά για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να παρέχουν πολλές θέσεις εργασίας και ε, να παράγουν πλούτο για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ και πολλές από αυτές είναι νεοφυείς επιχειρήσεις μάλιστα. Οπότε το σχέδιο γνωμοδότησης λέει ότι χρειάζονται έξυπνα συστήματα χρηματοδότησης που να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Και τέλος, χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, η συγκήτρια λέει ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια καλή γνωμοδότηση από πλευράς Επιτροπής Μεταφορών και η γνωμοδότηση έχει γραφτεί με τρόπο που να λάβει υπόψη της αυτά που λέμε ήτρε και να μην μπορεί να τα παραγνωρίσει, να τα άγνοησει. Ευχαριστώ πολύ. Σταματώ εδώ εξ ονόματος όλα αυτά της Κιζίνε μαϊσνε. Ευχαριστούμε κύριε Τέλιτσκα. Ο κύριος Μαρινέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και ευχαριστούμε και την εισηγήτρια για τις ιδέες στο σχέδιο γνωδότησης. Θέλω και εγώ να προσθέσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισάγει στην πρόταση του επόμενου πολιτείου του δημοσιονομικού πλαισίου χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση της αστυνομικής πολιτικής και των νέων δορυφόρων. Το νέο δορυφορικό σύστημα που μπορεί να εξυπηρετήσει και τις μεταφορές. Αυτό θα είναι σημαντικό ώστε στο μέλλον να καλύψουμε μελλοντικέ ανάγκες και χρηματοδότηση για να λειτουργούν τα διάφορα συστήματα. Επίσης, για τις μεταφορές το έγκνος θα πρέπει να καλύπτει όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες γωνιές που δεν καλύπτονται από το έγνος και θα πρέπει να προβλεφθεί και για το βιομηχανικό κλάδο μια πλήρης διασύνδεση με το έγνος, διότι μισά από τα αεροδρόμια χρησιμοποιούν το σύστημα προς στιγμή. Η Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί προτάσεις Ε, και στα πλαίσια της στρατηγικής μαζί να βρούμε λύσεις, νομοθετικές λύσεις, ώστε να πιέσουμε το βιομηχανικό κλάδο και τους διάφορες παρυφές της βιομηχανικής παραγωγής να χρησιμοποιήσουν την σχετική τεχνολογία. Διότι όταν βλέπουμε τους ευφυείς δρόμους λόγω χάρη, στους ευφυείς δρόμους καταφέραμε να το προβλέψουμε αυτό για τα αυτοκίνητα μέσω του γκαλιλαίου. Όμως ε, πρέπει να συνεχίσουμε. και να προβλεφθούν δέκτες για τον Γαλιλαίο από όλους τους φορείς που ασχολούνται σε αυτές, που σε αυτόν τον κλάδο και για τον Global Trekking. Διότι αυτή τη στιγμή η συχνότητα του BNB έχει κατοχυρωθεί Ξέρουμε ότι αυτή, αυτός ο εντοπισμός, το tracking, καλύπτει ένα μέρος μόνο του ενέργειου χώρου και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορεί να βελτιώσουν αυτές οι πρωτοβουλίες με πρόβλεψη για την καινοτομία στο διάστημα και για το μέλλον. Εάν θέλουμε να είμαστε διαστημική δύναμη η Ευρώπη, πρέπει κάτι να κάνουμε και την έρευνα. Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστούμε κυρία Μάστρα για την γνωμοδότηση αυτή και πράγματι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μία έκρηξη νέων δυνατοτήτων, νέων προτάσεων που θα έχουν να κάνουν και με τη χωροταξία, να έχουμε στοιχεία σε σχέση με την κινητικότητα των πόλεων, τις ε, εκπομπές, τη γεωργία, τις μεταφορές, αλλά και το έψι έχουμε και το κλάδο όμως πρέπει να ακούσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την καινοτομία, ιδίως στον χώρο του διαστήματος, θέλουμε ε, την ad hoc κατάλληλη ε, χρηματοδότηση για την πρόθεση τέτοιων έργων. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας και να στηρίξουμε νέα μοντέλα. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Έχουμε το ιστορικό ε, εκτοξευτεί με τους Αριάν αλλά και άλλους ε, επαναχρησιμοποιούμενες, ε, επαναχρησιμοποιούμενες εκτοξευτήρες. Μπορεί να μην είναι ότι καλύτερο, αλλά υπάρχουν τεχνολογία και υπάρχουν και κάποιες άλλες τεχνολογίες λιγότερο ψοκίνδυνες αλλά μπορούν να χρηματοδοτηθούν όπως μικρές ε, οι δορυφόροι, ε, οι μικροί που δεν χρειάζονται πολύ καύσιμο, αλλά έχουν περισσότερη ασφάλεια και αξιοπιστία. Πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε. Κρούν ε, τα τύμπανα του πολέμου κάποιοι στην... Ε, χτυπούν μάλλον τα τύμπανα του πολέμου κάποιοι και πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να περασπιζόμαστε την πολιτική του διαστήματο. Θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι και επίση θα πρέπει και στον τομέα των μεταφορών σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση και διάθεση των αποτελεσμάτων, να, να προωθήσουμε αυτές τις πτυχές. Είχαν, ε, είχε στοιχεία και ορίζον 2020 για το διάστημα. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνα έχει διαγράψει αυτά τα στοιχεία, δεν θα έπρεπε. Πρέπει να επανέλθουν στο πρόγραμμα, κατά την άποψή μου. Ό,τι έχει να κάνει με μεγαλύτερη αυτονομία, ασφάλεια, παλήθευση δεδομένων, δεδοφορικών δεδομένων, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Επίσης, θέλω να στηρίξω και τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών, όχι μόνο ε, οργανισμού για το Διάστημα, αλλά και το οργανισμό Άμυνα ε, και όλων των άλλων φορέων συνεργασία και οργανισμών που ε, έχουν κάθε συμφέρον να διευρυνθούν και προς άλλα κράτη-μέλη που δεν έχουν δορυφορικές δυνατότητες για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Να υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία και να μαθαίνουμε από τον άλλον. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φώστερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω την Κεζίνε Μάισνερ για την έκθεσή της. Πολύ πλόκος ο τομέας ε, το διάστημα. Ήμουν συντάκτρια γνωμήτης για την πρώτη χρονιά του NSSS στην Επιτροπή Ήτρε. Είχαμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε τον Καλείο. Τότε ήρθα και εγώ στο Κοινοβούλιο και βλέποντας τη διαδρομή που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια είναι φανταστικό πόσο προχωρήσαμε και σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Επίσης είναι σημαντικό το ότι η Γαλλία διατήρησε τις δυνατότητε εκτόξευσης όταν στη δεκαετία του 70 αποφάσισε το Ηνωμένο Βασίλειο να ε, αποσυρθεί, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί αυτό. Πολύ σωστά τα λέγε Αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς, ε, τον εντοπισμό, για ε, τις μεταφορές, ε, για να έχουμε πιο ακριβή ε, εντοπισμό, GPS, tracking, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά και άλλα ωφέλη με αυτά τα προγράμματα είχαμε. Ανθρωπιστικά ζητήματα, πάλι μπορούμε να βοηθήσουμε, να εντοπίσουμε και να δούμε πού συμβαίνουν διάφορα πράγματα στον πλανήτη μας. Ε, η συγγήτρια θα έχει ε, την υποστήριξη όλων. Πιστεύω ότι δεν είναι ένα θέμα που θα μας διχάσει, ανάλογα με τόση ποια πολιτική ομάδα ανήκουμε. Είναι μια απλή γνωμοδότηση, πολύ ξεκάθαρη και νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην ε, έκθεση της Καθήλυνα Αρμόδιας Επιτροπής με πολύ θετικό τρόπο ένα προσωπικό σχόλιο. Όταν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα βγει από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο. Σα το λέω για να το ξέρετε, γιατί η βιομηχανία του διαστήματο δεν είναι ευρωπαϊκή αμυγό, πολύ ευρύτερη και είναι καλό αυτό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Και κάποια από τα προγράμματα θα είναι κοινοπαραξίε στο μέλλον, όπω παραδείγματο χάρη όταν μπούμε στη φάση τη εφαρμογή, υλοποίηση. Είναι σημαντικό και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση, κατάλληλες διαδικασίες. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ και την κυρία Φώστερ. Θα μιλήσω κι εγώ ως συνεισηγήτρια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ για την πρότασή της. Συμφωνώ απόλυτα με τις διαπιστώσεις της, όμως το βασικό μήνυμα στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ διαστημικού προγράμματος και καινοτομία στις μεταφορές. Θα σας δώσω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Είτε πρόκειται για το EDRS, αυτούς τους δορυφόρους ε, που μας, δημιουργούν, ε, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δεδομένα σε τροχιά, ροή, βασική ροή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο παντού ε, στον κόσμο, είναι το πρώτο παράδειγμα, είτε το δεύτερο παράδειγμα πρόκειται για το πρόγραμμα Galileo, που θα δώσει ε, την ε, υπηρεσία γεωγραφικού εντοπισμού με ακρίβεια ε, του ενός μέτρου στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να έχουμε πάρα πολλές καινοτομίες στο μέτρο μεταφορών. Τα συζητούμε συχνά στην Επιτροπή μας, τα συνδεδεμένα οχήματα, τα αυτόνομα οχήματα κτλ. Αν θέλουμε η διαστημική τεχνολογία και τα εργαλεία της να υπηρετούν την καινοτομία, και την βιομηχανική αλλαγή στις μεταφορές θα πρέπει διάφοροι τομείς να επικοινωνούν και να έχουν μια κοινή στρατηγική. Είναι ε, χέρι-χέρι αυτά τα δύο. Καλή κλίμακα για να έχουμε τα στρατηγικά τεστ, γιατί είμαστε και από τους χρηματοδότες του ΕΣ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική στρατηγική συντονισμένη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης φορέων της και οργανισμών της. Θα είναι πραγματικά σημαντικό να το πετύχουμε. Θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες. Ελπίζω να μπορέσω να εκπροσωπήσω τη βιομηχανία αναφέροντας και τα αιτήματα της βιομηχανίας ε, με τις τροπολογίες μας. Γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, τα απορρίμματα, τα διαστημικά απόβλητα. Κανείς δεν το έχει αναφέρει αυτό το θέμα τεράστιο όγκο διαστημικών αποβλήτων. Δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε, δεν ξέρουμε τι απογίνονται αυτά τα απόβλητα. Άρα δεν έχουμε μόνο το θέμα της διαστημικής πρόοδου και τεχνολογίας ε, έτσι, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε με αυτά τα απόβλητα. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί με την πυρηνική ενέργεια, ξέρουμε παραδείγματος, τα πυρηνικά απόβλητα είναι μια καταστροφή, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Τα έχουμε ε, θάψει ε, στο υπέδαφος προς το παρόν, αλλά ε, θα πρέπει να δούμε μια οριστική λύση πρέπει να βρούμε. Βλέπω ότι ο κύριος Τέλιτσκα έχει σηκώσει το χέρι του. Ε, θα συνεχίσω λοιπόν. Ίσως απαντήστε και στο ερώτημά μου ε, μετά. Ο κύριος Ρικέ. να απαντήσω στο ερώτημά σας κυρία Πρόεδρε, όλα τα απόβλητα ε, παρακολουθούνται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν δύο οργανισμοί, ο ένας είναι αμερικανικός και μάλιστα λεπτομέρειες κάτω του εκατοστού. Τις παρακολουθούν πάρα πολύ στενά και υπάρχει και μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ε, να εκτοξευθούν ε, δορυφόροι, πειραματικοί, που να καθαρίζουν ε, και ακόμα και τα πιο μικρά απόβλητα, σαν τα μηχανήματα που μαζεύουν τα ψίχουλα. Είναι πάρα πολύ λεπτό αυτό το θέμα. Ένα λεπτό μικρό σχόλιο. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά τα όσα υπόθηκαν. Βέβαια, πάντα λέμε τι θα μπορούν να κάνουν για τις μεταφορές αυτές τις πρωτοβουλίες στο διάστημα, με ένα εξαντλητικό κατάλογο, τι μπορούμε να περιμένουμε από δεδομένα, ε, ε, τον ε, γεωγραφικό ε, εντοπισμό, μεταφορά δεδομένων για την εφοδιαστική και τις μεταφορές. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει το διάστημα. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι η πρόσβαση στο διάστημα είναι και αυτή από μόνη της ε, στοιχείο συστατικό των μεταφορών και το θεωρώ πολύ αφύσικο να μην το αναφέρουμε εδώ ως προτεραιότητα. Βεβαίως η ίδια η πρόσβαση στο διάστημα είναι μεταφορά, με μέσα μεταφοράς. Ε, και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο. Εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει ότι το διάστημα είναι κάτι που έχει να κάνει με την κυριαρχία. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, υπάρχουν ζητήματα αμυντικά και βεβαίω προβλήματα κυριαρχίας, πολιτικής ε, για την μεταφορά και τις μεταφορές και όχι μόνο. Έχουμε να ανησυχούμε πάρα πολύ επίσης ε, για τη συνέχιση των προγραμμάτων ε, εκτόξευσης. Ε, αυτή τη στιγμή είναι τριετή, είναι τετραετή. Δεν υπάρχει ορίζοντας χρονικός για τη χρηματοδότηση και έχουν κάνει προσπάθειες η Γαλλία και η Γερμανία για το πρόγραμμα Αριάν 6 και άλλα, αλλά δεν έχουμε μέσο μακροπρόθεσμα κανένα σχέδιο για την εκτόξευση δορυφόρων. Και δεν έχουμε εστίαση για την επαναχρησιμοποίηση των δορυφόρων. Είναι πάλι πολύ εύθραυστη, ευαίσθητη ε, αυτή η διάσταση και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να έχει ε, σημεία εκτόξευσης. Ε, η Αριάν 6, εντάξει πάνω κάτω καλύπτεται, αλλά η επόμενη γενιά είναι τελείως ακάλυπτη, δεν υπάρχει καμία προοπτική για το μέλλον και θα πρέπει από τώρα να ασχολούμαστε. Eh και βεβαίως ε, θα υπάρξουν ε, πτήσεις επανδρομένες ε, πολιτικής και όχι στρατιωτικές και στη στρατόσφαιρα ή κάτω από τη στρατόσφαιρα. Αυτά λοιπόν το διάστημα δεν είναι για μας τόσο πολύ η παροχή υπηρεσιών. Είναι μεταφορές και το διάστημα. Και θα πρέπει και εμείς λίγο να αναλάβουμε τα ενία. Γιατί κάπου το έχουμε αφήσει στη μοίρα του, ακόμα και αν είναι αρμόδια επί της ουσίας η Επιτροπή Βιομηχανίας Ήτρε. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε και να καταφέρουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια πρόταση ε, εγγράφου εργασίας. Γιατί το διάστημα δεν είναι κάτι το οποίο προγραμματίζεται 2, 3, 4 χρόνια. Η Ευρώπη πού είναι σε αυτή την ιστορία, πούσα έχουμε και μερίδιο στην αγορά, αλλά θα το χάσουμε αν συνεχίσουμε έτσι. Θα μας ξεπεράσουν οι πάντες στην επόμενη δεκαετία. Δηλαδή θα είμαστε ανύπαρκτοι σε λίγο και δεν θα έχουμε πρόσβαση στο διάστημα, άρα θα έχουμε χάσει και την κυριαρχία μας. Ευχαριστώ κύριε Ρίκη. Η κυρία Γοβονταλόν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια στο πρόσωπο του κυρίου Τελίτσκα για αυτή την τόσο πλήρη έκθεση που δείχνει πόση σύγκληση απόψεων υπάρχει από τους συναδέλφους εδώ σε αυτή την επιτροπή, επιτροπή για αυτό το τόσο βασικό θέμα. Δεν θα είμαι τόσο κατηγορηματική όσο ο κύριος Ρικέ, αλλά συμμερίζομαι πολλά από αυτά που είπε. Δηλαδή η διαστημική πολιτική της Ευρώπης εγγράφεται σε ένα τοπίο πολύ σαφές υπό, υπό χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών διαστημικών πόρων και του σκληρού ανταγωνισμού σε διεθνέ επίπεδο που απειλούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε αυτή την αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση πρέπει να στοχεύσει διαφορετικά σημεία, αλλά όταν ε, ακούω τι διάφορε παρεμβάσει των συναδέλφων εκ των προτέρων, καθησυχάζομαι. Η Επιτροπή μα μπορεί να λάβει σαφέστερη θέση υπέρ των ε, ρυθμιστικών προβλέψεων για να υπάρχει συμβατότητα διάφορων εγκαταστάσεων μεταφορών με τον Γαλιλαίο και προκειμένου να προβλέψουμε την εξέλιξη των ε, υποδομών που μπορεί να ε, αναπτυχθούν πολύ γρήγορα, όπω τα μη παντρωμένα αεροσκάφη και τα ευφύ αυτοκίνητα. Πρέπει επίση να κοιτάξουμε και τι κομπέ αερίων του θερμοκηπίου και το εξοδού του άνθρακα από τι μεταφορέ. Επίση, θα πρέπει να κοιτάξουμε να ε, μην βελτιώσουμε απλώ την ανταγωνιστικότητα των ξένων επιχειρήσεων ε, στην αγορά των δορυφόρων, όπω ε, τόνισε και ο κ. Ρικέ. όλε οι χώρε τη θεσμική του αγορά την έχουν προστατεύσει με συγκεκριμένε ρήτρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει προτίμηση στι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Έτσι, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλους ε, παραγωγούς ε, του εξωτερικού που επιδοτούνται αδρά ε, για την εκτόξευση Ευρωπαίων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δορυφόρων όπω ο Γαλιλαίο ή ο Κοπέρνικος. Θα πρέπει και εμεί λοιπόν να δώσουμε μια προτίμηση για του Ευρωπαίου παραγωγού στα πλαίσια της θέσης τροχιά των δορυφόρων που ανήκουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, η στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς της πολιτικής διαστήματος. Είμαστε στην ευχάριστη θέση και την ευτυχή να έχουμε ίδιοι όλες τις ε, γεωστρατηγικές ε, προϋποθέσεις για να στείλουμε, να εκτοξεύσουμε δορυφόρους και πύραυλους. Έχουμε ε, το κουρού στη Γαλλική Γουιάννα, υπάρχει το ΚΑΠ ε, που το οποίο είμαστε μέσα ανεξάρτητοι για να στείλουμε τους πυράβλους, ούτε εξαρτώμαστε από τον Μπαϊκονούρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι τεχνολογίες γενικά, τονίστηκε αυτό, έχουν οριμάσει και μάλιστα έχουμε τους πρώτους καρπούς. Ο Γαλιλαίο ε, γνώρισε πολλές κριτικές, ήταν τεράστιο πρόβλημα να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και από τα 8 δισεκατομμύρια που δόθηκαν πρόσθεσαν άλλο ένα δι στα κράτη-μέλη. Βρέθηκαν τα χρήματα όμως και το πρόγραμμα τώρα βρίσκεται, στο, έχει βάλει το δρόμο του και μπορούμε να έχουμε ένα Global Navigation Satellite System, το GNSS. Και έχουμε και ξεχωριστό ευρωπαϊκό οργανισμό με έδρα την Πράγα. Και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κύριος Τέλιτσκα. Πήγαμε ε, αποστολή στην Πράγα, ε, η Επιτροπή μας, και ε, μάθαμε ενδιαφέροντα πράγματα από τον εκεί διευθυντή. Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής ακόμα. Ας πούμε στην ασφάλεια των πτήσεων μας έδειξε ξεκάθαρα και ο Διευθυντής πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα και πώς ε, ε, είναι τα διάφορα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου στην Ευρώπη και πώς μπορούν να υποσυρθούν αυτά ή στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ακριβώς σε κάποια στενά. Ε, όταν είναι πολύ στενά ε, κάποια περάσματα και διασταυρώνονται δεξαμενόπλια όπως ε, κάποια θέματα που αφορούν την Ρωσική Ομοσπονδία ή ακόμα και στο Βόσπορο όταν έχουμε συνθήκες ομίχλης πολύ ισχυρών ανέμων καταιγίδων κλπ. Είναι μια ιστορία που πρέπει να τη συζητήσουμε πολύ σοβαρά στρατηγικά. Λοιπόν, να αφήσουμε της μικροδιαμάχης και ε, φιλονικής για το ποιο θα μαζεύει τα τέλη, τα διόδια κτλ. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε. Κάτι που δεν θα έπρεπε καν να υφίσταται. Όποιος πάει στη τσεχική δημοκρατία, στην Αυστρία, ξέρω εγώ, στη Γερμανία στο μέλλον, θα του κολλάνε ένα σήμα, μια βινιέτα. Στην, στην Ελβετία μπορώ να το φανταστώ, αλλά θα μπορούσαμε κι εμείς να το συμπεριλάβουμε αυτό. Υπάρχουν μεγάλοι πάροχοι που μαζεύουν τα χρήματα από τα διόδια. Το Στράντα είναι στην Ιταλία, στη Γαλλία Ντομινίκ και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, η Μπουίγκ. Όλοι αυτοί να χρησιμοποιήσουν ένα όμιλο όπως είναι η Airbus και άλλοι και να ε, πάρουν και τους μικρούς μαζί τους. Και να είναι ξεκάθαρα ότι ε, το, τα διόδια θα είναι σχετικά με, το, με τη συγκεκριμένη διαδρομή, με το συγκεκριμένο κράτος, να τα συλλέγει κάποιος και να κάνει και ε, το λογαριασμό. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει. Και κάτι που μας έκανε τεράστια εντύπωση, το GPS που το χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα κάνουν στο μέλλον οι Αμερικανοί, έχουν αρχίσει να στέλνουν και πειρά στη Συρία. Ούτε τι θα κάνουν οι Ρώσοι. Μπορούν από τη μία στιγμή στην άλλη να μας πούνε τέρμα το GPS, δεν θα χρησιμοποιείτε τους δικούς μας δορυφόρους. Άρα θα πρέπει εμείς το συντομότερο να το έχουμε έτοιμο να λειτουργήσει. Και αυτό το ευρωπαϊκό GPS, αυτό μας είπε ο Διευθυντής του Οργανισμού στην Πράγα, θα το έχουμε και ε, θα το φέρουμε σε ένα smartphone ή Android, αλλά η Apple θα μας το μπλοκάρει αν το μπλοκάρουν οι Αμερικανοί, αλλά μπορεί να το κάνει το Samsung. Και κάθε Ευρωπαίος να έχει μια τέτοια εφαρμογή στο τηλέφωνο του δωρεάν GPS, που είναι και πολύ πιο ακριβές κατά τα άλλα, συμπλήν 20 εκατοστά σε σχέση με το Αμερικάνικο. Και θα είναι και μια ευρωπαϊκή ταυτοποίηση, ε, θα ταυτίζεται ο κάθε Ευρωπαίος, θα έχει ευρωπαϊκή συνείδηση ότι εγώ είμαι Ευρωπαίος και έχω το ευρωπαϊκό σύστημα. Θα συμμετέχει η Βρετανία. Τα είπε Τζάκ, και εσύ Φώστερ ότι τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα συμμετέχετε και αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούν. Θα ακούσουμε για λίγα λεπτά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Λεπχενιέ, που είστε. Δεν είμαι κύρια όμως γιατί και Λεπκρενή είναι σε μια παράλληλη επιτροπή και συζητά το ίδιο θέμα, το θέμα της πολιτικής του διαστήματος, μου να την αντικαταστήσω. Θα σας το δώσω μετά το λόγο, ε, κύριε Τέλισκα Παρακαλώ, Επιτροπή. Ναι, θα τα πω αγγλικά όμως. Πρώτα απ' όλα να πω ότι καλωσορίζουμε την γνωμοδότηση και την υποστήριξη που εκφράσατε σήμερα στα σχολιά σας. Με την έγκριση και την εφαρμογή της στρατηγικής του διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο τα πλονεκτήματα της, ε, του διαστήματος τα φέρει στη γη για προστέμενη αξία τόσο για την οικονομία και την κοινωνία εν γέννη. Το είπατε και πολύ ότι οι μεταφορές είναι ένας τομέας κλειδί που μπορεί να ωφέλει μάλλα από τις θεσμικές εφαρμογές και νομίζω ότι είναι προφανείς και σημαντικές οι συνέργειες. Το είπατε και πολύ, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για κάποια από τα προγράμματα που έχουμε ήδη δρομολογήσει. Τον Καλλιλέο το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε και ένα δεύτερο σύστημα, το έγνος. Ένα περιφερειακό σύστημα που μεγεθύνει το, το σήμα ε, του GPS από το 2011 να ε, παραμείνω λίγο στο έκνος. Οι επιδόσεις αυτής της υπηρεσίας ε, ήταν εξαιρετικές. Το 2016 ήταν μια από τις καλύτερες του χρονιές. Ο κ. Μαρινέσκου όμως πολύ σωστά είπε ότι δεν έχει καλυφθεί επαρκώς όλη η επιφάνεια που θα θέλαμε και το δουλεύουμε το θέμα. Το 2016 το καλοκαίρι βελτιώσαμε τις υπηρεσίε, προσθέσαμε και περισσότερες υπηρεσίε. υπηρεσίες. Γενικά την τελευταία διετία έχουμε 12 δορυφόρου, έχουμε 8 σε τροχιά και τώρα είμαστε στα επόμενα βήματα. Να ολοκληρώσουμε την, ε, το όλο στερέωμα, αν θέλετε, για τι εκτοξεύσεις. Θα ήθελα τώρα να πω κάτι για το πρόγραμμα Κοπέρνικους που ίσως σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει των μεταφορών. Είναι ένα ενωσιακό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την παρατήρηση με κάποια άλλα στοιχεία για την επιτήρηση της γης. Έχουμε ήδη έξι υπηρεσίες ε, για το θαλάσσιο περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, την παρακολουθήση του κλίματος, ε, διαχείριση πηγόντων υπουργουσών ε, καταστάσεων, ασφάλεια κτλ. Το Κοπέρνικος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και για την ασφαλή ναυσιπλοεία, δίνοντας προφορίες, χάρη για την αρκτική, περιβαλλοντικές πληροφορίες κτλ. κτλ. Ένα τρίτο θέμα είναι μελέτη αντικτύπου για μια πιθανή πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τις ε, κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες που μπορεί να έχει εφαρμογές στη τη κυκλοφορίας, στον εντοπισμό, μπορεί να διευκολύνει και τα συστήματα ε, αυτόνομης ε, αυτοκινούμενων ε, ή τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων και ας πω και δύο λόγια για την αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα. Πολύ αναφέρεται στη στρατηγική του διαστήματος, λέμε ξεκάθαρα ότι έχουμε τη φιλοδοξία να βελτιώσουμε την αυτονομία της Ευρώπης στο διάστημα με ασφαλή ανεξάρτητη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στη στρατηγική μας περιγράφουμε κάποιες δράσεις που θέλουμε να αναλάβουμε προς το σκοπό αυτό. Τέλος. Σε σχέση με τα δικά σας σχόλια, νομίζω ότι αρκετοί είπατε ότι κάτι πρέπει να γίνει με την, ε, το μέρη της αγοράς ε, που θέλουμε να αυξηθεί, Γαλιλαίο κτλ. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Στη στρατηγική του διαστήματος Λέμε ότι η Κομισιόν θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβανομένων και ρυθμιστικών μέτρων όταν θεωρούνται ευεργετικά και δικαιολογούνται για αύξηση του μεριδίου του Γκαλιλαίου σε τομέα όπως κινητή τηλεφωνία, κρίσιμες υποδομές, αεροπορία. Άρα βλέπετε ότι το βλέπουμε, το βλέπουμε, μας απασχολεί και για την κινητή τηλεφωνία. Θα ολοκληρώσω δίνοντάς σας θετικές ειδήσει. Υπάρχουν ε, μεγάλη παραγωγή που έχουν ε, και η Samsung μεταξύ αυτών ε, βγάλει σε κυκλοφορία τηλέφωνα που δουλεύουν με δορυφορική τεχνολογία. Φυσικά και περιμένουμε να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Τέλιτσκα που του υποσχέθηκα θα του ξαναδώσω το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που στήριξαν την Κεζίνε και εξέφρασαν καλά λόγια για την ε, γνωμοδότησή της. Θα αντιστά, διαβιβάσω όλα αυτά τα θετικά σχόλια. Σε ό,τι αφορά ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις. Να απαντήσω σε μερικά από αυτά τα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στρατηγική του διαστήματο. Εξίσου σημαντικό όμω είναι, σε οποιαδήποτε άλλη στρατηγική που θα έχουμε στο μέλλον, να περιλαμβάνεται μια σκέψη σχετικά με τις ε, δυνατότητες μας, ε, τις διαστημικές δυνατότητες, Γκαλέο, Κοπέρνικους, Έγνος και ούτω καθεξής. Την υποδομή την έχουμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είμαστε μεταξύ των πρωταγωνιστών. Είμαστε σε καλή θέση. Ποιο είναι το πρόβλημα είναι ποιε είναι οι ευκαιρίε και δυνατότητε και από τη μία και ποιο είναι ο πραγματικό κόσμο από την άλλη. Το είπε και η πρόεδρο όταν μίλησε για τη διασύνδεση των διαστημικών τεχνολογιών με τι μεταφορέ και την καινοτομία συγκεκριμένα. Και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τι αφορέ, έχει να κάνει και με πολλού άλλου τόμου. Όταν πήγαμε στην Πράγα και επισκεφθήκαμε τον Γαλιλαίο, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψη. Αλλά ήταν ενδιαφέρον ότι δεν παίρναμε πάντοτε και όλες τις απαντήσεις που δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό, μια διαφορά μεταξύ ε, αφενός ημών και των ε, οργανισμών της Ένωσης και το τι μπορεί να γίνει. Ε, ποιοι τι κάνουν οι νεοφείς επιχειρήσεις, ποιοι παρέχουν τις υπηρεσίες, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. ώστε και η γνωμοδότηση της Γκεζίνε να περιλάβει κάποιο σχετικό σχόλιο. Ε, μεταφορά της μάλλον μεταφορά πραγματικότητας στις υποδομές. Αυτό είναι κάτι σημαντικό επίσης. Και πράγματι έχουμε το θέμα με τα απόβλητα. Έχουμε και την νομοθεσία και την κυκλική οικονομία όμως. Είναι το ίδιο με αυτό που είπα για τη στρατηγική του διαστήματος. Αμφίδρομο αυτό. Το ίδιο και η κυκλική οικονομία. Θα έχουμε τώρα τη βάση, θα έχουμε τα εργαλεία για να δώσουμε όθηση στη διαστημική τεχνολογία, όχι μόνο την ανακυκλώσιμη, αλλά που θα είναι και ε, μέσα στην κυκλική οικονομία. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε, δίνοντας κίνητρα. Και με την νομοθεσία που πέρασε στην Ολομέλεια, νομίζω ότι δίνουμε κίνητρα. Τρεις, τέσσερις παρατηρήσεις, παραδείγματος του κ. Μαρινέσκου, για ε, την ε, κυρία Μάισνερ προορίζονταν τα σχόλια, οπότε δεν θεωρώ εγώ ότι μπορώ να την καταστήσω και να απαντήσω εκ μέρους της. Αλλά θα τη διαβεβάσω ότι η μεγάλη πλειονότητα των σχόλων ήταν θετικά. Σας ευχαριστούμε κυρία Τελίντσκα. Έχετε ένα λεπτό κυρία Γελασέντερ. Ναι, ένα λεπτό για να απαντήσω για το θέμα των αποβλήτων στο διάστημα. Στις κάτω χώρες υπάρχει ένα αντίστοιχο κέντρο που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, στην ΕΣΑ, και μας έδειξαν ότι υπάρχουν έργα ακριβώς για την αποκομιδή των ε, διαστημικών απορριμμάτων. Κάτι θα κάνουν, θα ρίξουν ένα δίχτυ με το δορυφόρο και τα μαζεύουν ε, τα απόβλητα αυτά και τα γεννάνε πίσω. Ε, είναι κάτι σαν ένα καλάμι για ψάρεμα ή ένα δίχτυ για ψάρεμα, μια απόχη, τα μαζεύουν. Ε, βλέπω ότι σας ανησυχεί αυτό και πραγματικά το φροντίζουν, μην νομίζετε. Καλά, θα παρακολουθούμε στενά το θέμα αυτό των αποβλήτων. Δεν ξέρουμε καθόλου τι μπορεί να περιέχουν, οπότε αν ξανάρχονται στην ξηρά, ξηρά, εκτός μικροφώνου η απάντηση. Θα το παρακολουθούμε στενά. Θα το παρακολουθούμε στενά. Δεν θέλουμε να γίνει σκουπιδόντε νεκέ στο διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τελίντσκα. Ευχαριστούμε που εκπροσωπήσατε την κυρία Μάισνερ και που δώσατε ένα σύνολο απαντήσεων τόσο καλών στους συναδέλφους. Σας ενημερώνω ότι η προθεσμία για την υποβολή των είναι 19 Απριλίου, 12 το μεσημέρι τότε λίγη. 19 Απριλίου, 12 το μεσημέρι, δηλαδή σύντομα. Λοιπόν, τελευταίο σημείο. Ε, Έλεγχο. Παρουσίαση από την Επιτροπή του σχεδίου κατά εξουσιοδότηση πράξη για την έγκριση και αναθεώρηση τεχνικών πατεγραφών για τη διαλειτουργικότητα. Ο λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Ζούστ για 6 με 7 λεπτά το πολύ. Θα τα καταφέρετε? Τέλεια. Πολύ ωραία. Έχετε το λόγο. Πολύ σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το όντι θα σας παρουσιάσω την κατεξουσιοδότηση πράξη για τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργικότητα βασική διάταξη που δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο το γνωρίζει πολύ καλά η Επιτροπή σας πιστεύω. Έχει δύο πυλώνες. Το πιο σημαντικό αυτό που θα τώρα είναι ο τεχνικό, ο οποίο εγκρίθηκε στι 15 Ιουνίου πέρσι. Και θα γνωρίζετε το συνολικό πλαίσιο του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια ενιαία σιδηροδρομική περιοχή στην Ευρώπη με άρση των αναπομεινάντων φραγμών για να βελτιωθούν οι μεταφορέ μεταξύ των κάτω μελών και να δοθούν περισσότερες ευκαιρίε στις επιχειρήσει και του φορεί του κλάδου αυτού. Αλλά επίσης νέες υπηρεσίε και για τους επιβάτε και για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Κάτι που εξυπηρετεί του στόχου τη διάλειτουργικότητα, και επίση την επιδίωξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ω μέρο λοιπόν του τεχνικού πυλώνα, ε, προβλέπουμε και επιδιώκουμε μεγάλη απλούστευση όλου του ρυθμιστικού πλαισίου. Όπου εκεί θέλουμε να περιορίσουμε το διοικητικό κόστο και οι κατασκευαστέ, η παραγωγή, να μπορούν ανά την Ευρώπη και να αναπτύσσουν ε, την πώληση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα σημαντικό στοιχείο του τέταρτου συνδρομικού πακέτου είναι η άρση των εθνικών κανόνων εφόσον χρειαστεί. Χιλιάδες εθνικών κανόνων θα καταργηθούν μέσα από τη θεματική προσέγγιση. Υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία, ε, στοιχεία κλειδιά του τεχνικού πυλώνα, που είναι ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για την πιστοποίηση και την βεβαίωση ασφάλειας ξέρουμε ότι θα υπάρχει πια μια ενιαία θηρίδα ώστε να είναι ευθυνότερε οι διαδικασίε και συντονισμένη η διαδικασία πιστοποίηση. Όλο ιδιαίτερα αλλά όχι μόνο, για τι διασυνοριακέ υπηρεσίε. Η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με τον οργανισμό για να ετοιμάσει την υλοποίηση του τέταρτου σιδηροδρομικού πακέτου με τι ανάλογε μεθοδολογίε για να υπάρχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά και βεβαιώσει ασφάλεια, ο έλεγχο των ε, οχημάτων και αμαξοστοιχειών, το τροχιολικό και το καθεξής. Ε, όλες αυτές οι τεχνικέ υποδιαγραφέ για τη λειτουργικότητα δεν είναι ένα νέο στοιχείο ενό σιδηροδρομικού πακέτου, αλλά είναι αυτό που χρειάζεται διαρκή επικαιροποίηση και ενημέρωση ώστε να αντικατοπτρίζεται η τεχνική πρόοδο και όπου οι τεχνικέ περιγραφέ λαμβάνουν μεγαλύτερη σημασία, είναι εκεί που το, ο νέο οργανισμό σιδηροδρόμων θα πρέπει να δώσει τη δική του αδειοδότηση στο μέλλον. Ω προ τη συνεννόηση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 5 τη Οδηγία για τη Λειτουργικότητα, Οδηγία 2016-7 το άρθρο 5 ε, προβλέπει τη δυνατότητα για την Επιτροπή να εγκρίνει κατά εξουσιοδότηση ε, πράξη για την επικαιροποίηση αυτών των τεχνικών προδιαγραφών τη λειτουργικότητα. Αυτή την κατεξουσιοδότηση πράξη συζητούμε σήμερα. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτή τη εξουσιοδότηση πράξη είναι ότι πρέπει να εγκριθεί τώρα, πριν τι μελλοντικέ αναθεωρήσει ε, των τεχνικών προδιαγραφών τη λειτουργικότητα. Στο παρελθόν τα πρότυπα εγκρίνονταν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς ένα ε, πριτανεύον νομοθετικό πλαίσιο της βασικής οδηγίας. Τώρα πρέπει πρώτα να εγκριθεί η κατεξοδότηση πράξη για να δοθεί η δυνατότητα επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, προτεί εγκριθεί ε, με τη σειρά τη αυτή η νέα εκδοχή των τεχνικών προδιαγραφών. Έτσι, έχουμε μια ευκαιρία για να υπάρξει συνοχή μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητα και να είμαστε βέβαια ότι η υλοποίησή του είναι συνεκτική, συνεχή και να γνωρίζετε κι εσεί ε, κάθε στάδιο τη διαδικασία ω συνομοθέτε, αλλά το ίδιο και οι ενδιαφερόμενοι. Για το τι επιδιώκουμε συνολικά με τι τεχνικέ περιγραφέ και πώ μπορούμε να καθοδηγήσουμε τι συζητήσει για τι μελλοντικέ μα ανάγκε στο επίπεδο των τεχνικών περιγραφών και λειτουργικότητα. Μόλι εγκριθεί η κατεξουδότηση πράξη, που όπω είπα καλό θα να γίνει γοργά, θα γίνει η βάση και συγκεκριμένου στόχου που θα συνδεθούν με κάθε μια από τι τεχνικέ περιγραφέ ξεχωριστά. Αυτέ με τη σειρά του θα εγκριθούν στο μέλλον βάσει των συστημών συστάσεων που θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Οργανισμό των Σιδηροδρόμων. Οι ίδιε οι τεχνικέ προδιαγραφέ θα θεσπιστούν ε, με τη σειρά του, θα εκφραστούν μάλλον ε, σε τη πράξη βάσει του άρθρου 51.3 και τι ε, διαδικασίε εξέταση που προβλέπει ο κανονισμό. Για την τωρινή κατάσταση των τεχνικών προδιαγραφών έχουν περάσει από τι διαβουλεύσει με τον Οργανισμό των Σιδηροδρόμων πέρσι τον Ιούνιο, από τον Ιούνιο στον Αύγουστο. Έπειτα πέρασε μια μακρά περίπτωση εξέταση από την ομάδα εμπειρογνωμών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολλά πηγενέλα, με μια ακρόαση τον Γενάρη φέτο, όπου προσκλήθηκε το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι παραστήκατε σε αυτή την ακρόαση και μια περίοδο διαβουλεύσεων και πάλι μετά με 350 σχόλια τουλάχιστον ως τώρα, τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη και η τελική περίοδος για τις τελικέ απαντήσει τελικές και αποκρίσεις είναι ως τις 17 Απριλίου. Τρέχει τώρα. Μόλι ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινηθεί γοργά για την έγκριση τη πράξη, ώστε να ξεκινήσει και η περίοδο για να μπορούν να προβάλλουν ένσταση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Πάντω, σύντομα, η δομή τη πράξη. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια αρχικά άρθρα όπου έχουμε προσπαθήσει να ξεκαθαρίσουμε θέματα γενικού ενδιαφέροντο για όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, ιδίω για τις γενικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, απαιτήσεις να αξιολογείται το κόστος και ωφέλεια και ούτω καθεξής. Και πέραν αυτών υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα που καλύπτουν κάθε μια από τις 11 τεχνικές προδιαγραφές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για κάθε μια από αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Μερικά σημαντικά στοιχεία που πρέπει να σημειώσουμε και τα οποία αναφέρονται στην ΚΕΠ οι αλλαγές που προκύπτουν από το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και η ανάγκη συνοχής, η ανάγκη μεταβατικών περιόδων, το θέμα των πιστοποιητικών, τη ισχύω των πιστοποιητικών, την γίνεται όταν οι του επικαιροποιηθούν τι καθεστώς θα έχουν βάσει, των ισχυουσών του πουδού, πώς θα ακολουθήσουμε τα υποσυστήματα για συγκεκριμένα ε, οχήματα ε, ως μέρος της, μέρος της ανάλυσης και της μελλοντική ανάλυσης για τις εξελισσόμενες του πουδού, οριζόντια ζητήματα, η καινοτομία, οι προεκτάσεις της, στην ε, μετατόπιση προς τους συνδροδρομικές μεταφορές. Ξέρετε ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε την καινοτομία στο τομέα των συνδροδρόμων. Εάν δεν υπάρξει καινοτομία είναι σαφές ε, ότι δεν θα πρέπει αυτό να μείνει εκτός κανονισμού. Η ψηφιοποίηση, ή υπηρεσία πληροφορίας, και όλα τα υπόλοιπα συστήματα και δίκτυα που μας ενδιαφέρουν. Θα σταματήσω εδώ και αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστω. Είναι μαζί και ο ε, ειδικό που ήταν υπεύθυνο για τις υπομετεύσεις γύρω από το πακέτο, οπότε είναι εδώ και αν χρειάζεται κάποια ειδική ερώτηση να σας απαντήσει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσω τώρα τις ερωτήσεις. Κύριε Βαντενκάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε πολλές τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, και τέτοια θέματα λέμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτό ξαναπέστωλε, λέει κράμα. Ε, η καταξιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χαίρουν και μεγάλης προσοχής και εκτίμησης και είναι προσωπική μου γνώμη αυτό. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, πώς ε, Αναπτύστε μια κατεξοδότηση πράξη. Ο καθένας θέλει να ασχοληθεί με αυτή και με τις λεπτομέρειες στην κατάρτιση. Αλλά στην εφαρμογή τι γίνεται. Ξέρω ότι είναι ίσως πολύ νωρίς. Αλλά στις διαπραγματεύσεις για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο υπήρχαν κάποια κράτη-μέλη που ε, ακόμα εφήρμοζαν το δεύτερο πακέτο για τους σιδηροδρόμους. Ερωτώ λοιπόν, τι γίνεται με την εφαρμογή, ωραία όλα αυτά στη θεωρία και υπάρχει διαφορά μεταξύ κρατών μελών και σιδηροδρομικών οργανισμών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υποδομών. Γιατί υποθέτω ότι η κατεξοδότηση πράξη αυτή αφορά και τους οργανισμούς σιδηροδρόμων και τους διαχειριστές ε, των δικτύων και των υποδομών. Αυτή είναι η ερώτησή μου και θα παρακαλούσα να με διαφωτίσετε. Κύριε Κράμερ, εσείς. Ναι, η δική μου ερώτηση πηγαίνει προφανώς προς την ίδια κατεύθυνση. Στο τέταρτο σιδηροδομικό πακέτο αγωνιστήκαμε σκληρά να γίνουν κατεξουδότηση πράξη και να μην μας παρακάμψουν ότι είναι όλα τα τεχνικά και χαίρεται το Κοινοβούλιο να μην συμμετέχετε. Ε, ε, αν συγκριθούμε με σιδηροδρομικούς οργανισμούς, εμείς είμαστε πραγματικά ευρωπαϊκοί ενώ ε, ανεξαρτήτως χώρας οι οργανισμοί των σιδηροδρόμων είναι ε, οι τελευταίες ε, εθνικιστικές αρχές, κοιτάνε τη δουλειά τους και δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την Ευρώπη. Ήταν πολύ σκληρή λοιπόν η μάχη που δώσαμε, αλλά πετύχαμε να γίνει εξουσιοδότηση νομική πράξη. Δηλαδή ενημερωνόμαστε, εμείς αποφασίζουμε αν είναι τεχνικό το θέμα ή πολιτικό το εκάστοτε και μπορείτε να ποντάρετε και να προσβεύετε και στη δική μας υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν θα ξεχάσω τι είχε γίνει στο ERTMS που είπαμε ότι η συνδρομική αρχή θα πρέπει να έχει την τελευταία λέξη πόσο τα αγωνίστηκαν κράτη-μέλη εναντίον του. Που έλεγαν όλα καλά ήταν. Ενώ είχαμε αποφασίσει πριν από 12 χρόνια ότι το θέλουν το ERTMS, αλλά να είναι μια συγκεκριμένη βάση ε, συμβατή. Και έχουμε 10.000 χιλιόμετρα με ε, ε, ράγες, αλλά ούτε μία μηχανή ε, τρένου που να μπορεί να τη διανύσει αυτό το διάστημα. Και στο τρίτο πακέτο, στο τεχνικό πυλώνα, ε, συνεργαστήκαμε πολύ καλά οι συντονιστέ. Εγώ ανέκαθεν έλεγα στου Γερμανού, έχετε χάσει χρόνο και χρήμα 10 χρόνια και θα συνεχιστεί. Αν δεν μαθαίνετε ούτε από τα λάθη σα, πώ θα διαμορφώσετε το μέλλον. Τώρα έρχεται η ΕΡΑ, η Ευρωπαϊκή ε, ε, Σιδηροδρομική Αρχή. Ε, ωραία, αλλά πότε θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Όλα είναι ωραία στα λόγια και στους νόμους και στη διατύπωση, αλλά η κάθε χώρα μετά βγαίνει και κάνει τα δικά της. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα το επιβάλλεται αυτό. Όταν λέει ο ένας το Α και άλλο στο Β. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, όχι να μου. Ποια είναι η χρονική στιγμή, πότε θα συμφωνήσουν, αν δεν συμφωνήσουν τι θα γίνει, θα αποφασίσει η ΙΕΡΑ, θα αποφασίσετε εσεί, με το Κοινοβούλιο Ρήμεν των κρατών μελών. Πώ γίνεται αυτό, Πώ θέλετε να τα εφαρμόσετε όλα αυτά, για να μην έχουμε και άλλε ολιγορίε και χρονοτριβέ και εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε του στόχου μα ρεαλιστικά και ε, σε εύλογο χρόνο προς όφελο τη Ευρώπης και όχι οποιοδήποτε κράτο μέλο. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Ο κύριο Δελή. Uh, uh, ναι. Κάποιε ερωτήσει λόγω χάρη. Έχω κάποιο, κάποια δυσκολία με τι ασαφεί ε, διατυπώσεις. Φαντάζομαι ότι δεν είμαι μόνο όπω είπε και ο συντονιστή μα, ο διάβολο βρίσκεται στι λεπτομέρειε. Όντω, είναι πολλέ οι λεπτομέρειε σε ένα τέτοιο πλαίσιο, στο πλαίσιο που μα δώσατε το γενικό. Και λόγω χάρη το άρθρο 6 αυτού του πράγματο, αυτή τη κατεξουδότηση απόφαση τέλο πάντων, μιλάει για πραγματικό έλεγχο από τι μεταφορέ εμπορευμάτων. Ε, πραγματικό θόρυβο από τι μεταφορέ εμπορευμάτων. Δεν λέτε ποια θα είναι η προσέγγιση σα ακριβώ παρόλο που γνωρίζουμε ότι έχετε κάποια κράτη που είναι, υπάρχουν κάποια κράτη που είναι πολύ πιο αυστηρά, αλλά επί εκεί και κάποια κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που έχουν πολύ παλιό τροχαίο υλικό και πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του θορύβου που προκαλεί. Το άλλο θέμα που έχει να κάνει με το άρθρο 14 και την επισήμανση και την επισήμανση, κάτι που ήταν θέμα διακυβέρνησης για το τέταρτο συνδρομικό πακέτο. Τα εισιτήρια ε, για το τέλος της διαδρομής. Εδώ θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να αναλάβει το δικό του μερίδιο από αυτήν την ε, διαδικασία πριν ληφθεί μια τελική απόφαση. Και για το άρθρο 10, τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Σημαντικό θέμα. Έχουμε πάνω από 30.000 σιδηροδρομικούς σταθμούς, πολύ ψηλά σκαλοπάτια, και πολύ δύσκολη πρόσβαση για όσους βρίσκονται σε ένα παιδικό καροτσάκι ή έχουν οποιαδήποτε άλλη δυσκολία κίνηση. Όμως, για να βελτιωθούν τα πράγματα χρειάζεται πολύ χρήμα και χρόνος και κόπος. Η δική σας η πράξη, όταν τέλος πάντων περατωθεί, λαμβάνει υπόψη και αυτές τις παραμέτρους χρήμα και χρόνο. Πρόεδρος, και εγώ είχα εγγραφεί, διότι αυτό που σας ζωτούμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμερα, είναι πώς θα αναλάβετε δράση και αν ναι, αν σκοπεύετε να αναλάβετε δράση, πότε. Το έθιξε κάπως ο κύριος Ντελή. Θέλω και εγώ λοιπόν να σταθώ στο άρθρο 14 εδάφιο 6 της της πράξης. Νομίζω ότι είναι ε, το θέμα της άμεσης έκδοσης εισιτηρίων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα. Όπως λέει και η Οδηγία 2016, 2370, το τα πληροφόρηση για την έκδοση εισιτηρίων θα πρέπει ε, να λαμβάνει υπόψη του στην αγορά της λύσεις της διασυνοριακής πολυδιαλογικής παροχής υπηρεσιών. Στα σιδηροδρομικά θέλουμε ένα τέτοιο σύστημα με μη διακριτική μεταχείριση και με τρόπο διαλειτουργικό. Θέλουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορεί κανείς να σχεδιάσει τα ταξίδια του, τις μετακινήσεις του και την αγορά εισιτηρίων να είναι απλά και θέλουμε τα συστήματα αυτά να μην προκαλούν διακριτική μεταχείριση ε, ή ε, αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή όσων θέλουν να τηρήσουν το απόρριτο των εμπορικών πληροφοριών και ταυτόχρονα την προστασία, μάλλον το σεβασμό των καλών ανταγωνισμού. Τέλος πάντων, η τον ανταγωνισμο μεταξυ των σιδηροδρομικων επιχειρησεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να βεβαιωθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο και την υλοποίηση αυτών των σημείων. Και ε, πρέπει να μας υποβάλει κάποια στιγμή πραγματικές νομοθετικές προτάσεις. Οπότε, το ερώτημα, λίγο πολύ, είναι πολύ απλό. Έχετε πρωτοβουλίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα. Και αν ναι, πότε θα τις δούμε. Κύριε Κράμερ, θέλετε περώτηση. 30 δευτερόλεπτα. Ναι, πολύ σύντομα. Αυτό με τις πληροφορίες πανευρωπαϊκά για τα εισιτήρια, για τις πληροφορίες. Στα τρένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Παγκοσμίω βλέπει όλες τις πληροφορίε. Είτε είναι 27 χώρες, 30. Ε, και έρχονται και είναι οι συνδρομικοί οργανισμοί ότι είναι απόρριτα αυτά, ότι είναι μυστικά, ότι είναι χεμήθεια, τι ίδιε είναι αυτέ. Και του είπαμε έχετε τρία χρόνια να το κάνετε, Έλλειω θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το κάνει. Θέλετε να απαντήσετε σε ένα-δύο λεπτά. Αλλιώς συγκεκριμένα να μας απαντήσετε με mail. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Βαντενκάμπ για την νομοθεσία και πώς θα εξασφαλίσουμε την σωστή μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Δεν αφορά βέβαια αυστηρά την κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά συνολικά όλες τις διατάξεις του πακέτου. Έχουμε συνεργαστεί με τα κρατημέλη τους, έχουμε πει ότι μέσω της Επιτροπής που ασχολείται με τα αριθμιστικά ζητήματα θα τους δώσουμε λεπτομερείς οδηγίες για τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, ιδίως εκεί που υπάρχουν κάποια ζητήματα που είναι τόσο ξεκάθαρα για όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουν γρήγορα και ομοιόμορφα να μεταφέρουν όλα τα κράτη-μέλη στην εθνική τους νομοθεσία της Διατάξης. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν πώς θα μεταφέρουν την νομοθεσία στο δίκαιο, μπορεί να μην τη μεταφέρουν σωστά, μπορεί να τη μεταφέρουν πιο αργά. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Έρχομαι στον κύριο Κράμερ για την συνεκτική προσέγγιση ή μη. Κάτι καινούριο, πολύ σημαντικό στο τέταρτο πακέτο είναι ότι δεν βασιζόμαστε απλά και μόνο στα κράτη-μέλη για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και για την χορήγηση αδειών με βάση εθνικούς κανόνες που θα πρέπει να συνάδουν με το βεβαϊκό πλαίσιο. Δίνουμε τη δυνατότητα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, αν θέλουν, να έρθουν στο σιδηροδρομικό οργανισμό για τα πιστοποιητικά ασφαλείας και για τις εγκρίσεις, για τις Και με τη διαδικασία αυτή βέβαια ο οργανισμός θα εφαρμόζει με ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την Ευρώπη τους δικούς μας κανόνες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι έτσι ορισμένα από τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν θα εξαλειφθούν, τέλο πάντων θα μειωθούν στο ελάχιστο. Αυτό προσπαθούμε, δηλαδή να καταργήσουμε στο δυνατόν του εθνικούς κανόνες και με τις μελλοντικέ βελτιώσεις ε, στις ε, ε, τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας νομίζουμε ότι θα διορθώσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και τις αποκλήσει που είχαμε ανάλογα με τα κρατημέλη. Τρία ζητήματα για την χορύπανση, την έκδοση εισιτήριων μέχρι τελικό προορισμό και την προστασμότητα. Για το πρώτο θέμα χορύπανση, πολύ ε, ε, σωστά το είπατε και υπάρχει πλαίσιο. Αυτό παρέχει η ε, τεχνική προδιαγραφή, και συζητήσαμε και με τα κατημέλη και με τον Οργανισμό Συνδεδρόμου για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πολύ λεπτό αυτό ζήτημα για τους λόγους που κι εσείς οι ίδιοι έχετε εκθέσει, ώστε να είναι δυσανάλογα τα μέτρα. Να αντιμετωπίζουμε τις πολύ θεμητές ανησυχίες για την ε, υγεία. Δηλαδή δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου στις άλλες χώρες. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς νομίμως μπορούμε να προχωρήσουμε. και για αν χρειάζεται να γίνεται εκτροπή. Με τα TSI, με αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές, θα δούμε ε, αν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η προσέγγιση και με τις νέες ε, τεχνικές, ε, τεχνολογικές εξελίξεις που θα τις περιλάβουμε στην προδιαγραφή για να βρούμε σωστές λύσεις. Το through ticketing, η έκδοση δηλαδή με το τελικό προορισμό, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα με την προδιαγραφή. Εμείς θα σπίσουμε το τεχνικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τις ώρες, ε, για τις τιμές των κτλ. Η προδιαγραφή όμως από μόνη της δεν μπορεί να επιβάλλει σε δρομικές επιχειρήσεις να διαθέσουν σε τρίτους ε, την, να σε τη δυνατότητα πώλησης ε, εταιρεί, εισιτήριου. Εξαντλήσατε το χρόνο σας, λέει η Πρόεδρος. Εγώ θα ήθελα να δεσμευτείτε κύριε Φύς ότι θα μας στείλετε ιδίως για αυτό το θέμα της ε, έκδοσης εισιτηρίων και για τα άλλα θέματα που δεν απαντήσατε ένα email πολύ συγκεκριμένο. Διότι εμεί είμαστε νομοθέτες και είναι επίγουσα η σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διατυπώσει προτάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και μάρτυρες είναι όλοι οι συντονιστές. Κύριε Φύς, περιμένω με ανυπομονησία το mail με τις διευκρινήσεις, εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους βουλευτές, κυρίως τη λήξη τη συνεδρίαση οι συντονιστές 6 με 7 λεπτά από τώρα, ξανά εδώ, πάρτε και το καφεδάκι σας για να αντέξετε μέχρι τις 6.30. Τα λέμε σε 6-7 λεπτά.